Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σας μέρα. Θα έλεγα να εγκρίνουμε την μέσα διάταξη πρώτα. Εγκρίνεται πολύ ωραία. Έχω κάποιες σύντομες ανακοινώσεις να σας κάνω. 21 Νοεμβρίου 2017 ε, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, την εποπτεία scrutiny slot, θα το αφιερώσουμε στο PSD2, θα καλύψουμε όμως και το IFR. Το χρονοδιάγραμμα τώρα για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής το 2018 και τις συνεδριάσεων των συντονιστών ε, έχει εγκριθεί. Οι συντονιστές συμφώνησαν να λάβει η χώρα μια και τη συνεδρία της 11 Δεκεμβρίου 2017 στο Στρασβούργο για να συζητήσουμε το τραπεζικό πακέτο Είπαμε επίσης ότι θα χρησιμοποιήσουμε το υπάρχον πάνελ για τον ε, νομισματικό διάλογο ε, το 2018. Θα πρέπει να δώσουμε έγκαιρα και τις γραμμές ότι φορά τις δράσεις που πρέπει να λάβουμε λόγω της λήξης του υπάρχοντος πλαισίου. Σε ό,τι αφορά τώρα την ομάδα εργασίας ε, χρηματοπιστωτικής συνδρομής, οι συντονιστές συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα οικονομική διακυβέρνηση. Οι συντονιστέ συμφώνησαν να καλέσουν τον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ στην συνεδρίαση του, σε μια συνεδρίαση του 2018. επίση θα μα παρουσιάσει την ετήσια έκθεση του European Fiscal Board στι αρχέ του 2018. Σήμερα θα συζητήσουμε επίσης τη διαβούλευση τη ΕΚΤ για τα NPL, για τα ε, δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα. Και βεβαίω. θα μας μιλήσει και η κυρία Νούη. Υπάρχει το θέμα της συμμετοχής στην διαβούλευση. Στη συνέχεια έχουμε την δημόσια ακρόαση για τα ΠΕΠ. Ε, συμφωνήσαμε συντονιστές να καλέσουν πέντε εκπροσώπους, κάποιον από την Αμούντι, κάποιον από την Αλιάντς, από τα Ολλανδικά εξωτερικά Ταμεία, τον κύριο Μποέρι και έναν εκπρόσωπο της BEUC, BEUC. Θα πρέπει να έχουμε ισότιμη εκπροσώπηση των φίλων στον μέτρο του δυνατού εγκρίθηκε μια αιτήσια έκθεση από τους συντονιστές. Επίσης ε, υπάρχει και το αίτημα για τις, ε, τα ψηφίσματα 048-2017 που θα τεθεί στην επόμενη συνέντευξη των συντονιστών ως ε, θέμα και εξετάσαμε και το θέμα της εργασιών γύρω από το Brexit. Και τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω την Ντανιέλ Νουή, επικεφαλής της Εποπτικού Συμβουλίου ε, στην Ευρωπαϊκή Εταιρική Τράπεζα είναι η δεύτερη τακτική ακρόαση του 2017 όπως προβλεπόταν στον οργανισμό SSM και τη Διαθεσμική Συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα είχαμε ξαναπεί τον Ιούνιο του 2017. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που αφορούν τον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Τομέα αυτή τη στιγμή θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Φαντάζομαι χαίρομαι που είστε εδώ σήμερα και σας ευχαριστώ για αυτό. Έχουμε εντοπίσει δύο σημεία κυρίως. Πρώτα το περίφημο addendum για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το προπερασκευαστικό έργο στην ΕΚΤ ε, για την εποπτεία των ε, τραπεζών εν ώψη του Brexit. Σε ό,τι αφορά το addendum, γνωρίζετε ότι υπάρχει το θέμα των θεσμικών αλλαγών. Είχαμε και μια συζήτηση από αυτού κλεισμένου των θυρών. Το συζητήσαμε και σε επίπεδο Άλλωστε, η μείωση της ε, έκθεσης ε, των εκτιθυμένων δανείων τέλο πάντων, των εξυπηρετούμενων, είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό ότι μειώνεται, μειώνεται σημαντικά ε, το ποσοστό των μη εξυπηρετημένων δανείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στα κάτι μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο. Οι καθηγητέ γραμμέ του Μαρτίου λοιπόν του SSM από ό,τι φαίνεται είναι αποτελεσματικέ έω τώρα καθώ και τα μέτρα που έχουν παθεί σε εθνικό επίπεδο και σε τραπεζικό επίπεδο. Όμω το πρόβλημα δεν έχει ακόμα επιληθεί. Και όπω είπε πρόσφατα ο κύριο Δράγκη, χρειάζεται να γίνει μια κοινή προσπάθεια από τι τράπεζε, τι εποπτικέ αρχέ, τι ρυθμιστικέ αρχέ, τι εθνικέ αρχέ έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ε, όσο γίνεται πιο οργανωμένα. η Επιτροπή ΕΚΟΝ θέλει να συνεισφέρει επικοδομητικά και θετικά σε αυτήν την κοινή προσπάθεια. Και καλωσορίζω τα επιπλέον μέτρα που αναφέρονται στο σχέδιο δράσης που ενέκρινε το ΕΚΟΦΗΝ του Ιουλίου καθώς ε, και στην πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το νέο αντέντουμ ε, στις κριτές γραμμές του Μαρτίου που έθεσε προς διαβούλευση το SSM ε, σκοπεύει να αποτελέσει μέρος αυτής της κοινή προσπάθειας. Βεβαίως όμως ε, εδώ πάμε πέρα και από το Συμβούλιο και από την Κομισιόν και τις οδηγίες τους. Εμείς ε, ε, αναγνωρίζουμε ε, πλήρως τις εξουσίες, τις αρμοδιότητες του SSM για να επηρεάσει την πολιτική των τραπεζών για τα μη ξυπνούμενα δάνεια εντός όμως των ορίων που προβλέπονται. Υπάρχει μάλιστα συγκεκριμένη διατύπωση στην ανακοίνωση της Κομισιόν γι' αυτό. Είναι αυτή η αρμοδιότητα αλλά και καθήκον, υποχρέωση της εποπτικής αρχής. Ε, όσοι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή όμως το addendum πάει πέρα από τι αρμοδιότητες αυτές. Ε, οι αρμοδιότητες αφορούν τις τράπεζες, σαφώς, αμυγό. Εδώ αναφέρονται κάποιοι γενικοί κανόνες που αφορούν όλες τις τράπεζες και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω τη κατάλληλη τροποποίηση τη νομοθεσία για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τις αρμοδιότητες των συνομοθετών, ζητήσαμε επίσημη γνώμη από την νομική υπηρεσία, ε, τη δική μας, που έφτασε στο συμπέρασμα ότι η άσκηση των εξουσιών εποκτείας που έχουν αρμόδιες αρχές εξαρτάται από την επιμέρους κατάσταση, επιμέρους περίπτωση της κάθε τράπεζας που ε, και επιτρέπει μέτρα μόνο που αφορούν την εν λόγω τράπεζα το addendum όμως ε, εδώ προβλέπει επιπλέον υποχρεώσεις για τις τράπεζες που πάνε πέρα από το ρυθμιστικό πλαίσιο το υπάρχον. Η νομική υπηρεσία αποδεικνύει σαφώς με βάση την ομολογία πως ε, ο μηχανισμός συμμόρφωσης και εξήγησης και οι συγκεκριμένοι όροι σε ό,τι αφορά και τις εξαιρέσεις ε, για τη συμμόρφωση, σχέση με τη συμμόρφωση αυτή έχουν νομικές επιπτώσεις, έχουν νομικό αποτέλεσμα. Και αυτό ε, πάει πέρα από το άρθρο 3 ε, που προβλέπει να πάμε πέρα από το πλαίσιο. Διότι εδώ δημιουργούμε μια επιπλέον ουσιαστική υποχρέωση και αυτό αλλάζει, τις αλλάζει τον ρόλο της υποπτικής αρχής. Ε, δημιουργείται έτσι μια σύγχυση μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα που πρέπει να είναι σαφώς διακριτή. Ακόμα και στον τίτλο του αντέντου μου, το γεγονός ότι αναφερόμαστε ε, σε μία, ε, ένα μέτρο που μπορεί να πάρθει μόνο μέσω νομοθεσίας, περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Στα πλαίσια της συνεργασία και της συμφωνίας μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων, εμείς θέλουμε να συνεισφέρουμε ε, για να βελτιωθεί αυτό το αντέντουμ και να ευθυγραμμιστεί με τις αρμοδιότητες ε, των υποπτικών αρχών, δηλαδή πρώτα ε, αξιολόγηση που να αφορά αμυγός στις τράπεζες ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και στα πλαίσια του διαλόγου διαθεσμικά και όπου χρειαστεί επιπλέον μέτρα. Εμείς αναμένουμε να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση ελπίζουμε να υπάρχει μια ανοιχτή στάση και από το SSM, δηλαδή να είμαστε ανοιχτοί εννοούμε και σε αλλαγές, σε αλλαγές και του αντέντουμ, έτσι ώστε να αποφύγουμε ε, αντιπαράθεση αχρίαστη μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Τώρα υπάρχουν και άλλα σχόλια σε αφορά το περιεχόμενο. Ε, θα επανέλθω σε αυτά αργότερα όταν θα πάρω το λόγο. Όμως πριν δώσω το λόγο σε εσά, θα ήθελα να κάνω ακόμα δύο προσθήκες. Πρώτον, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε σαφέστερα ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των ροών ε, και των μετοχών. Εδώ μιλάμε για νέες ροές. Όπως είπε και η Κομισιόν και το Συμβούλιο, δεν πρέπει να υπάρχει εδώ καμία αναδρομικότητα. Αλλιώς θα συνειδητοποιήσουμε τις μετοχές, διότι θα ήταν αντιπαραγωγικό να, έχουμε, να, οδηγήσουμε, να οδηγηθούμε σε πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επίση, όλα τα δάνεια αποτελούν μέρο των κανόνων περί αναδρομικότητα. Η διαβούλευση που θα ολοκληρωθεί στι 8 Δεκεμβρίου και που στη συνέχεια θα τεθεί σε ισχύ 1η Ιανουαρίου, ε, αυτό το διάστημα είναι πολύ μικρό. Ελπίζουμε λοιπόν η SSM να δώσει αρκετό χρόνο στον εαυτό της να εξετάσει ε, τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης και ε, επίσης να μπορέσουν και οι τράπεζες να προετοιμαστούν εγκαίρως για αυτές τις νέες κατευθυντές γραμμές. Όπως και να έχουν τα πράγματα, μια μελέτη αντικτύπου ε, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για να δούμε ποιος θα είναι οι αυτών των μέτρων. Ευχαριστώ, Ντανιέλ. Σου δίνω το λόγο ευθύ αμέσω. Yes. Good Καλημέρα σας, καλημέρα πρόεδρε. Είναι χαρά μου να συζητήσω σήμερα τις εργασίες του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Τέσσερα τα θέματα που με ενδιαφέρουν σήμερα. Η αναθεώρηση του κανονισμού του SSM, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προπαρασκευές για το Brexit και τέλος τα αποτελέσματα ε, των ε, εποπτικών δοκιμασιών αντοχής για το 2017. Τώρα για τον κανονισμό του SSM, του ενιαίου μηχανισμού. Είναι θετικές οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον κανονισμό. Η αποτελεσματικότητα της εποπτείας της τραπεζικής βελτίωσε γενικότερα την κατάσταση στην περιοχή του ευρώ, στην ζώνη του ευρώ. Η αξιολόγηση είναι θετική λοιπόν, περιλαμβάνει φυσικά και ορισμένες δυνατότητες και προτάσεις βελτίωσης, τις οποίες εξετάζουμε προσεκτικά. Κάποιες από τις συστάσεις αυτές αναφέρονται στη λειτουργία του SSM γενικότερα και η πρακτική τους εφαρμογή θα έχει συνέπειες και σε επίπεδο λειτουργικό και σε επίπεδο νομικό και γι' αυτό η δική μας αξιολόγηση θέλει ακόμα κάποιο χρόνο. Να έλθω τώρα στα κόκκινα δάνεια, στα μη εξυπηρετούμενα είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει τα κέρδη, μειώνει μάλλον τα κέρδη των τραπεζών, κάτι το οποίο είναι προβληματικό σε μια θα έλεγα ε, περίοδο χαμηλής κερδοφορίας. Ταυτόχρονα είναι κάτι το οποίο ε, εμποδίζει την παροχή νέων δανείων στο παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας. Απέναντι σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η βελτίωση των ενεργών των τραπεζών είναι κάτι το οποίο ήταν ο βασικός μας στόχος από την αρχή που λειτουργήσαμε σαν SSM. Η προσπάθειά μας καλύπτει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα επίπεδα πιστοτικής δραστηριότητας. Στην Τραπεζική Ένωση οι τράπεζες δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται επί τη βάση της ε, εθνικότητάς τους, αν και διέπονται φυσικά από την εθνική νομοθεσία. Σαν ένα πρώτο βήμα δημοσιεύσαμε τις ε, ποιοτικέ συστάσεις NPL τον Μάρτιο του 2017 ζητήθηκε από τις τράπεζες να υιοθετήσουν ε, ρεαλιστικά και σίγουρα αξιόπιστα προγράμματα, φιλόδοξα προγράμματα για την αντιμετώπιση των NPL, των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τον τελευταίο χρόνο είδαμε μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα να κάνουν τεράστιες προσπάθειες για τη μείωση του στόκ των NPL στα οποία έχουν στο σύνολο της Ευρωζώνης. Υπήρξε λοιπόν μείωση ε, κατά 142 δις. Έφτασαν τώρα πλέον τα NPL σε 795 δις το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Φυσικά απαιτείται περαιτέρω δουλειά στον τομέα αυτό. Με βάση λοιπόν την συγκεκριμένη της εντολή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα <clears throat> θα πρέπει να προσπαθήσει σε προληπτικό επίπεδο να αντιμετωπίσει τους κινδύνους στο μέλλον μαθαίνοντας από την παλαιότερη εμπειρία. Από τότε που δημοσιεύσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές μας προς τις τράπεζες σχετικά με τα κόκκινα δάνεια, συνεχίζουμε την προσπάθεια λήψης περαιτέρω μέτρων αντιμετώπισης του θέματος. Πάντα ήμασταν πάρα πολύ διαφανείς. Ξεκινήσαμε τη διαβούλευση το Σεπτέμβριο του 2016 και ήδη ανακοινώσαμε ότι η προσπάθεια που κάνουμε σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια δεν θα ολοκληρωθεί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας μόνο στο στόκ των MPL που υπάρχουν σήμερα, αλλά θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα αποφύγουμε στο μέλλον μια σώρευση αντίστοιχη τέτοιου είδους μη εξυπηρετούμενων δανείων. Συνεπώς λοιπόν έφτασε η στιγμή να κάνουμε το επόμενο βήμα. Έχουμε σημαντικά ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες πλέον στην Ευρώπη, πρέπει να εκμεταλλευτούμε την όθηση αυτή, παίρνοντας μακροπρόθεσμα μέτρα, σε εποχές τις οποίες θα έλεγα ιδιαίτερα θετικές και πρόσφορες. Γι' αυτό λοιπόν εμείς συντάξαμε ε, μια πρόταση προσθήκης στην κατευθυντήριε στις κατευθυντήριες γραμμές NPL. Ξεκίνησε η διαβούλευση στις 4 Οκτωβρίου σχετικά με τα νέα NPL, όχι τα νέα δάνεια γενικά. Και εμείς θέλουμε να αποφύγουμε ακριβώς αυτό το οποίο είχε συμβεί στο παρελθόν και να μην υπάρξει περαιτέρω αύξηση των μη εξυπηρετούμενων στο μέλλον. Η πρόταση προσθήκης προτείνει ότι τα ακάλυπτα δάνεια θα καλυφθούν μετά από δύο χρόνια αυτή τη στιγμή χαρακτηριστούν ως ε, μη εξυπηρετούμενα. Για τα καλυμμένα θα πρέπει να υπάρξει μια πρόταση για 100% κάλυψη μετά από 7 χρόνια κατά τη διάρκεια της επταετίας αυτής έχουν ταξινομηθεί ως μη εξυπηρετούμενα. Και εμείς θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αυτή μετά από την Ιανουαρίου του 2018. Παρ' όλα αυτά πρόκειται για μια διαβούλευση, οπότε όλα μπορούν να αλλάξουν, ακόμα και οι χρονικές προσθεσμίες. Το θέμα έτσι και αλλιώς του χρονοδιαγράμματος είναι κάτι το οποίο μπορεί να επανεξεταστεί. Πάντως αυτό το αντέντομα αυτή η προσθήκη αυτή τη στιγμή υιοθετηθεί εντάσσεται στα πλαίσια των εποπτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι ένα μέσο α, του πυλώνα υπαριθμών 2 και απαιτεί να λαμβάνονται μέτρα μετά από κατά περίπτωση μελέτη και δεν θα υπάρχει κανένας αυτοματισμός εδώ. Η πρόταση προσθήκης απλά διευκρινίζει προς όφελος της διαφάνειας και της ισότητας ανάμεσα στα πιστοτικά ιδρύματα ποιες είναι οι εποπτικές μας προσδοκίες σε σχέση με την πιθανή δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων. Οι τράπεζες και γενικά τα πιστοτικά ιδρύματα ε, ζητήθηκε μάλλον από αυτές να μας δώσουν τις απόψεις τους για τις προτάσεις αυτές. Από τότε που δημιουργηθήκαμε είμαστε διαφανείς σε σχέση με τις προσδοκίες τις οποίες έχουμε εμείς, ακόμα και σε επίπεδο μη δεσμευτικών ποσοτικά ε, συστάσεων, σαν παράδειγμα η κατανομή των κερδών είναι μια σύσταση προς τις τράπεζες. Η ερμηνεία λοιπόν την οποία δίνουμε εμείς στην προτινόμενη αυτή ε, πρόταση παραρτήματος είναι ένα μέσο που ανήκει στον πυλώνα 2. Ε, και αυτό επιβεβαιώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο, τότε το SSM αντίστοιχα με άλλες εποπτικές αρχές στον κόσμο δεν θα είχε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το μέσο αυτό το τόσο σημαντικό για τα ευάλωτα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Όπως είπε επίσης και ο πρόεδρος του Eurogroup, υπήρχε γενικότερη υποστήριξη από πλευρά τη ομάδας στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πρόταση παραρτήματος είναι συμβατή επίσης και με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τα μη εξυπηρετούμενα. Το Συμβούλιο είπε ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στις τράπεζες για να αντιμετωπίσουν τα μη εξυπηρετούμενα ε, και ακριβώς οι προτάσεις μας ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση. Να σας υπογραμμίσω επίσης και να σας υπενθυμίσω ότι προς όφελος της διαφάνειας και για να υπάρξει πραγματικά σωστή συλλογή απόψεων από τους εμπλεκομένους δεν έχουμε πάρει παρά μία και μόνη απόφαση, να ξεκινήσουμε μία δημόσια διαβούλευση. Η διαβούλευση αυτή λοιπόν θα συνεχιστεί μέχρι την 8η Δεκεμβρίου του 2017 και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα επανεξετάσει όλα τα σχόλια τα οποία θα έχει λάβει πριν κάνει την τελική της πρόταση για την προσθήκη, για το αντέντουμ. Έρχομαι τώρα στις προετοιμασίες για τον Brexit. Από τότε που αποφάσισε το Ηνωμένο Βασίλειο να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, το SSM είναι σε συνεχή διάλογο με πολλές τράπεζες που επηρεάζονται από το Brexit. 50 τράπεζες ε, ήρθαν σε επαφή μαζί μας είτε απευθείας είτε μέσω των εθνικών εποπτικών αρχών, άπαξ αλλά και επανειλημμένα. Μερικές πολύ μεγάλες διεθνείς τράπεζες οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ευρώ μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν προγραμματίσει, έχουν προχωρήσει στον προγραμματισμό της αντιμετώπισης του θέματος. Κάποιες τράπεζες έχουν ζητήσει ε, τη διεύρυνση της αδειοδότησής τους που αξιολογούνται στην παρούσα φάση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές Πιστοτικές Αρχές. Πάντω, πάρα πολλέ τράπεζε καθυστερούν να πάρουν την τελική τους απόφαση για την αναδιάρθρωση των λειτουργιών τους, αφήνοντας τις επιλογές τους ανοιχτές. Αξιολογώντας τα σχέδια μεταφοράς των τραπεζών, είδαμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα. Ιδιαίτερα υπάρχει μια τάση να δημιουργούνται κενές περιεχομένου πιστοτικές εταιρείες στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξαρτώνται από υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά από το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει επίσης και τάση μεταφοράς τραπεζικών δραστηριοτήτων σε επενδυτικές εταιρείες τρίτων χωρών, εκτός δηλαδή ελέγχου του SSM και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ρυθμιστικής διαιτησίας. Εδώ λοιπόν εξαρτώμεθα από τους Ευρωπαίους νόμοθέτες να υπάρξουν οι απαιτούμενες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο. Σημαντικές λοιπόν τράπεζες της ζώνης ευρώ που έχουν δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζονται και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι προετοιμασίες αυτές και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τις πιστοτικές τράπεζες, τα πιστοτικά ιδρύματα συγγνώμη προς την κατεύθυνση αυτή. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει επίσης ε, και την ανάλυση της ε, ευαισθησίας ε, των τραπεζών στις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Όπως είπαμε, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα ανατράπεζα χρησιμοποιήθηκαν και για να λάβουμε αποφάσεις σε επίπεδο ΣΡΕΠ. E τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας. Τρεις βασικές σκέψεις, τρία συμπεράσματα βγαίνουν από αυτό. Πρώτον, η έκθεση στις διακυμάνσει των επιτοκίων φαίνεται αρκετά περιορισμένη. Κατά μέσο όρο, μια απότομη αύξηση του ύψου των επιτοκίων θα έχει θετικά αποτελέσματα στα κέρδη των τραπεζών και μια ελαφρά αρνητική, αν θέλετε, επίπτωση ε, στην πραγματική αξία των ενεργών της τράπεζας. Είναι σημαντικό να δούμε εδώ ότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης βρίσκονται σε διαφορετική μεταξύ τους κατάσταση κάτι το οποίο είναι παρηγορητικό αν θέλετε υπό το φως του κινδύνου της υπερβολικής συγκέντρωσης των προβλημάτων και των κινδύνων. Δεύτερον, σε σχέση με την αξιοπιστία των τραπεζών ε, που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε σχέση με τη συμπεριφορά των πελατών στο μέλλον. Σαν παράδειγμα, ε, το κόστος της λιανικής τραπεζικής δραστηριότητας θα παραμείνει σταθερό ακόμα και αν αυξηθούν τα επιτόκια. Όμως πολλές φορές τα σενάρια αυτά βασίζονται ε, σε μια λογική η οποία διαμορφώθηκε σε μια εποχή μείωσης των επιτοκίων και γι' αυτό τώρα τα πράγματα αλλάζουν με την πιθανή αύξηση. Γι' αυτό λοιπόν εμείς βρισκόμαστε σε διάλογο σε επίπεδο λεπτομέρεια σημαντικό με τις μεμονωμένες τράπεζες. Οι έλεγχοι τους οποίους κάναμε δείχνουν ότι έχουν κάνει σημαντικές προσπάθειες στον τομέα των παραγόγων για τα επιτόκια, όχι μόνο για να προχωρήσουν σε ένα σωστότερο hedging όπως θα το ανέμενε κανείς, αλλά και για να ε, μπορέσουν να καλύψουν καλύτερα τους ισολογισμούς τους. Το θέμα είναι λοιπόν να διαβεβαιώσουμε ε, το κοινό ότι η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί. Κλείνω τώρα τις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις εφόσον επιθυμείτε. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να έχετε την δυνατότητα να δώσετε περαιτέρω απαντήσεις σαν παράδειγμα τις δυνατότητες συμμόρφωσης ε, από πλευράς των πιστοτικών ιδρυμάτων, των οδηγιών που έχουν κυκλοφορήσει σε διάφορα επίπεδα. Είπατε ότι δεν υπάρχει αυτοματισμός και μόνο όταν γίνεται μία ανάλυση κατά περίπτωση είναι κάτι το οποίο προτείνει το κείμενό σας και αυτό είναι θετικό. Αυτά όλα σημαίνουν ότι τα πράγματα βελτιώνονται αλλά υπάρχει και περαιτέρω χώρος βελτίωσης. Πρώτος ο μιλητής ο κύριος Ροζάτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστούμε την κυρία Νοή για αυτήν την ε, συνοπτική παρουσίαση του παρατήματος της κατευθυντήρες γραμμές ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το πρώτο μου ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω ε, είναι, αφορά το μη χαρακτήρα, τη μη τραπεζικού χαρακτήρα πτυχή της, ε, αυτού του παρατήματος. Ε, δηλαδή δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο δεν είναι δεσμευτικό αυτό το, αυτή η πτυχή. Γιατί όταν εμείς διαβάζουμε αυτό το παράρτημα, διαπιστώνουμε ότι σίγουρα επιβάλλει ορισμένες υποχρεώσεις στα τραπεζικά ιδρύματα. Ε, ακούσαμε και την ε, άποψη της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου ε, η οποία μας είπε ότι έτσι όπως είναι διατυπωμένο αυτή τη στιγμή αυτό το παράτημα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό γιατί ο μηχανισμός δεν έχει κάποιες αρμοδιότητες σε αυτό το πλαίσιο. Δεύτερο ερώτημα. Θεωρείτε πως αυτές οι ποσοτικού χαρακτήρα διατάξεις θα μπορούσαν να έχουν ε, αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών, ε, το, τον, το ρυθμό του κύκλου των δραστηριοτήτων των τραπεζών σε περίπτωση που υπάρξει μια νέα κρίση. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση ε, τέτοιου είδου διατάξει δεν θα οδηγούσαν τελικά στην υποχρέωση τη τράπεζα να περάσουν σε υψηλή αποθεματοποίηση. Πράγμα το, βέβαια το οποίο θα είχε και, μια λυσιδωτή αντίδραση. Ε, στην οικονομία. Από εκεί και μετά, ε, ένα γενικότερο ερώτημα. Η Επιτροπή ε, πρόσφατα υιοθέτησε μια ανακοίνωση σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της Αμερικής Ένωσης και ζητάει από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν το ταχύτερο δυνατό κάποιες προτάσεις σε ό,τι αφορά τη μείωση του κινδύνου των τραπεζών και επίσης προτείνει κάποια βήματα σε ό,τι αφορά το, την υιοθέτηση ε, του European Deposit Insurance Scheme. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στο επίπεδο του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την έγκριση αυτών των βημάτων. Οπότε, ε, εσείς πώς θεωρείτε ότι θα μπορέσουμε τελικά να επιτύχουμε πρόοδο σε ό,τι αφορά αυτό το σύστημα, το European Insurance Deposit. Α Ε, ας ελπίσουμε ότι σημερινά η ακρόαση θα παράσει κάποιες διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά σημαντικά ζητήματα, όπως αναφέρθηκε ήδη και από τον ε, Πρόεδρο. Δεν θα ε, υπάρξουν αυτοματοποιημένες, ε, αυτοματοποιημένες Τώρα, απαντώντας στο, ταυτόχρονα και στο ερώτημα του Πρόεδρου, ναι, η δική μου αξιολόγηση είναι ότι ναι, το τρέχον κείμενο αναφέρει κάτι τέτοιο, αλλά όταν ακούω τόσους πολλούς να εκφράζουν κάποιες αμφιβολίες, τότε προφανώς διαπιστώνω ότι μπορεί να βελτιωθεί και πράγματι θα βελτιωθεί η διατύπωση που έχουμε εδώ. Ναι, και το να λέμε, να εξηγούμε καλύτερα, ίσως δεν είναι ο πιο εύστοχος για να χρησιμοποιήσουμε εδώ. Ας δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις σε αυτό το έγγραφο. Και από εκεί και μετά προφανώς θα τις λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας όλες ε, αυτές και τις νομικές, ε, νομικού χαρακτήρα συμβουλές που θα λάβουμε. Και αν ε, στα τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου δεν είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε πλήρως αυτά που μας έχετε προτείνει, τότε θα αποφασίσουμε ότι ναι, αρχε ιανουαριου Ιανουαρίου, 1η Ιανουαρίου δεν θα είναι η καλύτερη ημερομηνία για να ε, ξεκινήσουμε. Θα, προφανώς, θα προσπαθήσω προφανώ να πείσω τον ε, συνοντά μου, αλλά ε, σε κάθε περίπτωση ναι, θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, να δώσουμε περισσότερο χρόνο στον εαυτό μα για να λάβουμε σοβαρά υπόψη μα όλα αυτά τα σχόλια που θα έχουν υποβληθεί. Τώρα, αυτό το procyclical ε, effect, ε, αυτό το κίνδυνο δηλαδή να υπάρξει τέτοιο αντίκτυπο ε, που αναφέρατε, ε, ειλικρινά δεν νομίζω ότι υπάρχει ε, τέτοιο κίνδυνο. Ε, εντάξει, έχουμε κάποιου πολίτε που αντιμετωπίζουν προσωπικέ δυσκολίε στο επίπεδο τη ανεργία. Ναι, εκείνοι μπορεί να. σε εκείνους μπορεί να υπάρξει κάποιος αντικτυπός, αλλά αυτά που μας λένε τα στατιστικά στοιχεία μας ε, μας καταδεικνύει ότι βρισκόμαστε στην κατάλληλη φάση γιατί ακριβώς είναι καλύτερη οικονομική κατάσταση. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη βελτίωση της οικονομικής συγκυρίας. Θα ήταν πολύ δύσκολο δηλαδή για τις ε, ε, τράπεζες, την οικονομία και γενικά τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρεθούν στην επόμενη κρίση, γιατί ξέρουμε ότι κάποια στιγμή κάπου, δεν ξέρουμε πώς και πότε, αλλά θα υπάρξει στην ε, επόμενη κρίση. Δεν θέλουμε λοιπόν να δούμε ε, τις τράπεζές μας να αντιμετωπίζουν μια νέα κρίση ε, χωρίς να έχουν μάθει, αν θέλετε, τα διδάγματά τους από το παρελθόν. Σε ό,τι αφορά τώρα την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. όπως έχω πει επανειλημμένα, θεωρώ πως είναι κατάλληλη χρονική συγκυρία για να περάσουμε σε αυτήν την φάση δηλαδή της ολοκλήρωσης της Ένωσης. Αν πάρουμε για παράδειγμα το παράδειγμα της Banco Popular, αν δεν είχε αγοραστεί από την ε, Santander, αν δηλαδή αυτό δεν είχε αποδοθεί, ε, και η καταθέτες ε, δεν είχαν λάβει την αποζημίωσή τους, δεν είχε υπάρξει εποπτεία ε, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας, γνωρίζετε τι θα είχε συμβεί. Και στην Πορτογαλία, όπου είχαμε για παράδειγμα μια δημιουργία θηγατρική και όπου υπήρξε αποζημίωση των καταθετών, βλέπετε τι έγινε και τι επιτύχαμε σε αυτό το επίπεδο. Εγώ σημειώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει λάβει κάποιες πρωτοβουλίες για να προσπαθήσει ακριβώς να υπερκεράσει αυτό το πολιτικό αδιέξοδο που έχει προκύψει σε ό,τι αφορά την προώθηση αυτού του φακέλου της ε, ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και είμαι πεπισμένο ότι κινούμαστε προς την κατεύθυνση του πλήρους έντης όπως είχε δηλαδή ε, πρόταθεί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, γιατί και εγώ ε, θεωρώ πως αυτός θα πρέπει να παραμείνει ο βασικός στόχος και υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας των πιστωτών να προτιμούμε να επιτύχουμε αυτή την ένωση. Ο κύριος Ζάτη φαντάζομαι ότι εννοούσε στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο έτσι. Η έχει το λόγο. Ναι, Ευχαριστώ. Θα επανέλθω στον συνάδελφο Σίλβα Περέιρα στο θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σα ευχαριστώ για τι διευκρινήσει που δώσατε σχετικά με την ερμηνεία, ε, που, την αθασμένη από ό,τι φαίνεται, για τα περιεχόμενα του μου, Αυτό που θα πρέπει να διευκρινίσουμε ενδεχομένω είναι τη θέση σε, το θέμα τη θέση σε, ισχύος, σε ισχύ και ποια θα είναι η διαφορά μέσα στι ροέ και στα αποθέματα. Ε, μπορείτε να μας τα πείτε ίσως αυτά σήμερα, χωρίς να περιμένω αποτελέσματα της ε, διαβούλευσης. Θα ήταν ε, καλοδεχόμενη μια τέτοια πληροφορία. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο για τις ESA της Ένωσης της Εποπτικές, διότι μια από αυτές η EBA ε, εμπίπτει στις αρμοδιότητες σας, τις αρμοδιότητες της δικής σας ε, οργάνωσης. Πώς βλέπετε εσείς ε, την σχέση μεταξύ ρύθμισης και εποπτείας, έτσι όπως το προτείνει η Κομισιόν, πώς διαρθρώνεται η εργασία, των, οι εργασίες ε, του SSM και της EBA. Και ένα ερώτημα για τη μέθοδο που χρησιμοποιείται σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση μιας τράπεζας, ε, το κατά πόσο δηλαδή υπάρχει ρίσκο πτώχευσης ή όχι. Αναφερθήκα στην περίπτωση του Banco Popular. Ε, και βλέπουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο αξιολογήσατε αυτήν την πιθανότητα πτώχευσης ε, επηρεάζει την δυνατότητα κεφαλοποιήσεις μιας τράπεζας και το σύνολο της διαδικασίας ε, και έγινε μια ολόκληρη συζήτηση για το θέμα αυτό των συνθήκων εντός των οποίων λαμβάνει η χώρα αξιολόγηση. Είναι λοιπόν σημαντικό νομίζω να επανέλθουμε από αυτού. Σας ευχαριστώ επίσης για την αξιολόγηση ε, για το ίντις και την, για την υπενθύμηση ότι χρειαζόμαστε ένα πλήρες ε, ίντις τελικά ε, διότι από δική μας πλευράς η ανακοίνωση της Κομισιόν έτσι όπως το λέγουμε εμείς τουλάχιστον δεν συνεισφέρει σε αυτή την πλήρη εξασφάλιση και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να το διορθώσει αυτό. Ναι, να απαντήσω για το EBA και τα ESA γενικότερα. Ε, για την EBA να πω καταρχήν ότι ήταν κρίσιμη για να αναπτύξουμε το εγχειρίδιο για το μοναδικό κανόνα και τους σχετικούς κανόνες ε, χωρίς τους, τον ορισμό της ΕΜΠΑ για την έκθεση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα του 2014. Σίγουρα θα χρειαστούμε την EBA ε, για αυτό το εγχειρίδιο έτσι ώστε να υπάρχει μια συνέπεια σε ό,τι αφορά ε, τις ε, ίσες ευκαιρίες σε ρυθμιστικό επίπεδο, διότι αν δεν υπάρχει ρυθμιστικές κατευθύνσεις γραμμές ε, του EBA πρέπει να έχουμε νέα διαφορετικές ομάδες δικηγόρων, 19 μάλλον ομάδες δικηγόρων για να αναλύουμε το κάθε νομικό πλαίσιο. Αυτό δεν αποτελεί χρηστή διαχείριση, δεν αποτελεί αποτελεσματική εποπτεία. Έχουμε κάποιε επιφυλάξει ότι τι προτάσει για την EBA, διότι η EBA δεν είναι όπως η ΕΣΜΑ, δεν μπορεί να είναι η εποπτική αρχή για την ε, ενιαία κεφαλαία αγορά. Είναι κάπως διαφορετική η κατάσταση. Υπάρχει και ένας άλλος Ευρωπαίος επόπτης ε, πέρα από την Ιμπία. Οι προτάσεις όσο έχουν εδώ δημιουργούν μια σύγχυση ε, σε ό,τι αφορά τους ρυθμιστικούς και τους εποπτικούς κανόνες για το εκτελεστικό συμβούλιο της EBA. Εδώ έχει υποστεθεί μια επιπλέον έμεση εποπτεία στην πρόταση. Δεν είμαστε πεπισμένοι ιδιαίτερα για την πρόταση ό,τι αφορά τη συγκέντρωση του, του στρατηγικού προγραμματισμού στο εκτελεστικό διοικητικό συμβούλιο, γιατί αυτό δεν δίνει επαρκή ευελιξία στις αρμόδιε αρχέ για να αντιδράσουν όταν προκύπτουν ρίσκα ε, και κίνδυνοι κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού. Ε, Επίσης ε, συμφωνούμε με, με την υπάρχουσα κατάσταση σε ό,τι αφορά τα stress test. Αυτή η προσέγγιση ε, μέσω των, με, με, ευρω, με πανευρωπαϊκά stress test ε, υπό την εποπτεία και την έγκριση του, του Διοικητικού Συμβουλίου του EBA, αλλά δεν ξέρουμε αν πρέπει να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες γιατί για τέτοιες σταθεριότητες σε μια μικρή επιτροπή που δεν συμμετέχει στην άμεση εποπτεία. Διότι είναι μια δουλειά που έχει να κάνει με την εποπτεία. Όσοι έχουν τα πράγματα τώρα είναι τέλεια. Αν όμω ε, οδηγηθούμε ε, προς την κατεύθυνση που προτείνει η Κομισιόν, εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι σκόπιμο. Γενικότερα τώρα για τις αλλαγές σε επίπεδο διακυβέρνησης, εμείς καλωσορίζουμε ε, την προσπάθεια να έχουμε μια πιο ευρωπαϊκή εστίαση δεν είμαι βέβαιο ότι έχει δικαίωμα ψήφου πρόεδρο του EBA και που είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει νομίζω να εξεταστεί να μπορεί ο πρόεδρο του EBA να έχει δικαίωμα ψήφου, να έχει... διότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή φωνή. Επίση η ΕΚΤ δεν προβλέπει να συμμετάσχει στο εκλεστικό συμβούλιο ε, του EBA, παρότι είναι Ευρωπαϊκή Αρχή, η οποία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία σημαντικών θεσμών στα πλαίσια τη Ευρωζώνη. Αυτά είναι ζητήματα που μα απασχολούν. Σε ό,τι αφορά τώρα την ανακεφαλαιοποίηση, το τελευταίο που είπατε, εδώ το σημείο κλειδί, όπως ε, αναφέρεται άλλωστε στην νομοθεσία και τις διευκρινήσεις που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι αυτή η ανακεφαλαιοποίηση δεν πρέπει να καλύπτει ε, τις απόλυτες του παρελθόντος και πρέπει να οδηγήσει σε βιώσιμους, ε, βιώσιμα ε, θεσμικά όργανα μετά το τέλος της ανακεφαλοποίησης. Εγώ θεωρώ ότι οι κανόνες, το πλαίσιο, ε, ο, ο επιχειρησιακός χαρακτήρας του πλαισίου, όχι οι αρχές αυτές καθ' αυτές, θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω, θα πρέπει να υπάρξει μια ευθυγράμμιση, διότι είναι περίπλοκο. Ε, είναι μακροσκελές, κρατάει χρόνο και δεν είναι καλό να περιμένει μια τράπεζα πολύ καιρό ε, την απόφαση για την κεφαλοποίηση, γιατί υπάρχει αβεβαιότητα. Αυτό δεν είναι καλό ούτε για την τράπεζα, ούτε για του επενδυτέ, ούτε για του καταθέτε. Λειτουργεί πάντω το σύστημα, έχει δοκιμαστεί για μια σειρά από τράπεζε, αλλά κατά τη γνώμη μου θα ήταν καλύτερο να είναι λίγο πιο γρήγορη η διαδικασία να διευθυνθεί περισσότερο, η μεθοδολογία. Ευχαριστώ. Ashley Fox. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλημέρα κυρία Νούη. Έχω τέσσερα σύντομα ερωτήματα να θέσω. Πρώτον, ποια επίπτωση θα έχει το high leverage ratio τύπου 5% ε, στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής οικονομίας η οποία βεβαίως είναι σε ρυθμούς ανάπτυξης αλλά ε, σιγά σιγά. Δεύτερον, ε, υπάρχουν τα μορατόρια powers. Αυτό όμως μπορεί να έχει ε, και κάποιες επιπτώσεις μη ε, Μπορεί να υπάρξουν εκπρόσωποι τρίτων χωρών να χρησιμοποιήσουν, το, θα χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματα, ε, το δικαίωμα opt-out από τα πρωτόκολλα EFTA. Ε, στέλνεται επίσης ένα αρνητικό μήνυμα στην αγορά και αυτό ε, διακυβεύει την οικονομική σταθερότητα. Μια λύση δύο ημερών ε, ως προθεσμία δεν θα ήταν πιο κατάλληλη Τρίτον, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θεωρείται με την Σάντα Λούνε στην Φλαμανδή συνάδελφο προ την έκθεσή τη για την Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι τα κράτη-μέλη και οι ίδιε οι τράπεζε έχουν την πρώτη ευθύνη για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και τέταρτον, κάτι τελείω διαφορετικό τώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είπε ότι θέλει να εφαρμόσει ένα ευρωπαϊκό ε, hub για την fintech. Ε, πώς μπορεί να γίνει αυτό, διότι μπορεί να προκύψουν ζητήματα αδειοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. Well, you Γνωρίζετε ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της Βασιλείας 3 η Ευρώπη δεν ήταν πάρα πολύ υπέρ της ε, υψηλότερης χρήσης του level ε, ratio. Από την άλλη καλό θα ήταν να υπάρχουν διαφορετικά μέσα για την ε, προσμέτρηση των κεφαλαιοχικών αναγκών του κάθε, της κάθε τράπεζας. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες πηγαίνουν σχετικά καλά, πλησιάζουν τα επίπεδα απαιτήσεων και είμαστε στο 5,1 κατά μέσο όρο για τα σημαντικά τραπεζικά ιδρύματα. Πηγαίνουμε λοιπόν σχετικά καλά. Τώρα μη αναμενόμενες συνέπειες του μορατόριου, pre-resolution ή όχι. Κοιτάξτε, εμείς ε, το έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό με τους συναδέλφους και στο SRB και είχαν την τάση θα έλεγα πριν να εξετάσουμε και περιπτώσεις όπως την Banco Popular ότι ήταν ένα μέσο για τις... Uh, and uh, uh, Είναι ένα μέσο για να περάσουμε σε μια διατεταγμένη πρόβλεψη πτώχευσης κλεισίματος ε, της, ε, του Τραπεζικού Ιδρύματος. Από ό,τι φαίνεται θα σας πούν οι συνάδελφοί μου αν διαφωνούν, ότι το να υπάρξει ένα moratorium pre-resolution είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποφασίσει περισσότερο το SRB και όχι τόσο το SSM. Είναι πάντα δύσκολο να μπορέσει κανείς να ζητήσει το να κλείσει ας πούμε μια τραπέζα μέσα σε λίγες μέρες θα ήταν καλό για το SRB να περιμένει κανείς να περιμένουμε την Παρασκευή για να ανακοινώσουμε επίσημα ότι μία τράπεζα έχει πτωχεύσει. Να αποφύγουμε δηλαδή τέτοιου είδους ενέργειες στα μέσα της εβδομάδας. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να δούμε πότε θα κλείσουμε την τράπεζα, ποια είναι η καλύτερη στιγμή. Πάντως είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά ευαίσθητο, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφασίζεται σε σύντομες χρονικές προθεσμίες, αλλά θα πρέπει να υπάρχει περισσότερος χρόνος για να εξηγιάνουμε σε εισαγωγικά την τράπεζα. Αν ισχύει ένα τέτοιο μορατόριο δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε εμείς ο πρώτος πελάτης που φτάνει στην τράπεζα να εξυπηρετηθεί καλύτερα από αυτόν ο οποίος είναι δεύτερος. Αυτό είναι το θέμα της ισότητας της αντιμετώπισης των καταθετών ή των επενδυτών. Είπατε ότι η βασική ευθύνη ανήκει στα κράτη-μέλη. Κοιτάξτε, πράγματι ε, ε, το εποπτικό κομμάτι είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ένωσης ε, της Τραπεζικής. Υπάρχουν και άλλα θέματα όμως τα οποία ξεπερνούν το εποπτικό πεδίο, σαν παράδειγμα τα εθνικά νομοθετικά πλαίσια. Γι' αυτό ακριβώς μας πήρε πάρα πολύ χρόνο για να κάνουμε τις προτάσεις για τα εθνικά νομικά πλαίσια έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι πηγαίνει καλά σε κάποια τέτοια πλαίσια και μειώνει τα προβλήματα και τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Αλλά είναι σαφές όπως είπατε ότι ένα βασικό κομμάτι του προβλήματος είναι η αλλαγή του νομικού πλαισίου των νομικών διακανονιστικών ρυθμίσεων, των εθνικών διακανονιστικών ρυθμίσεων, κάτι το οποίο γίνεται. Ευχαριστώ Πρόεδρε. κύριο Σόμπο. Ευχαριστώ την κυρία Νουή η οποία έρχεται εδώ και μας ενημερώνει με τόσο σοφό τρόπο. Πρώτον, Nous parlons de l'union bancaire. Nous, nous la voulons, nous la désirons dans la zone euro. Εμείς θέλουμε να υπάρχει τραπεζική τράπεζα, γιατί αλλιώς θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει κάτι το πραγματικά ωφέλιμο για τους πληθυσμούς της Ευρώπης. Μήπως όμως de facto υπαναχωρεί Βλέπουμε ότι το Popolar αγοράστηκε από μια Ισπανική τράπεζα. Αν μιλήσουμε για τις δύο Ιταλικές τράπεζες, εξαγοράστηκαν από Ιταλικές τράπεζες. Ο αριθμός των διασύνοριακών ροών των τραπεζικών συναλλαγών, δηλαδή τραπεζικών ιδρυμάτων που εγκαθίσταται σε άλλες περιοχές της Ευρώπης κτλ. μειούται. Ε, είμαστε ε, μάρτυρες μιας επανεθνικοποίησης της πιστοτικής δραστηριότητας. Συμφωνείτε, σας απασχολεί αυτό. Δεύτερον, έντις. Θα συμφωνήσω με τους δύο προλαλήσαντες και θα προσθέσω τις ανησυχίες μου. Είπατε ότι είστε ικανοποιημένοι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεμπλόκαρε την κατάσταση. Ε, το πιστεύετε τώρα αυτό. Μήπως έχουμε να κάνουμε με μία νέα μικρή ε, κομπίνα έτσι ώστε να αποκρύψουμε την πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να κλείσουμε την ε, Τραπεζική Ένωση γιατί δεν υπάρχει ε, κοινή ανάληψη ευθύνη σε σχέση με την ανάληψη κινδύνων και την ανάληψη πρωτοβουλειών για την αξιολόγηση των κινδύνων. Θα συμφωνήσετε με αυτόν τον νέο ρυθμό ο οποίος υποθετικά επιβάλλεται γιατί ε, τώρα υπάρχει εμπιστοσύνη, αλλά μετά από πέντε χρόνια θα μας πούνε ότι ε, τώρα εντάξει αφού πάνε καλά τα πράγματα δεν χρειάζεται να επιμένουμε. Τώρα για τα α, ε, μη εξυπηρετούμενα, εγώ δεν α, ε, ομιλώ ως εκπρόσωπος μιας υπηρεσίας τραπεζικών συμβούλων. Εγώ κάνω λόμπι, αλλά κάνω λόμπι για τους Ευρωπαίους πολίτες και τους Ισπανούς κυρίως πολίτες που με εκλέγουν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το πώς θα το πετύχετε. Αυτό το οποίο πρέπει όμως να πετύχετε είναι να μην κινδυνεύουμε ε, να περάσουμε μια κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος όπως αυτή που βιώσατε. Ε, πράγματι σε σχέση με το στόκ, ας προσπαθήσουμε να το ρυθμίσουμε σωστά, αλλά και οι συναλλαγές στο μέλλον. Πρέπει να πάρουμε πραγματικά όλες τις πιθανές προφυλάξεις, γιατί όλες αυτές λειτουργούν αρνητικά για τον Ευρωπαίο πολίτη. Παρακαλώ οι ερωτήσεις σας να μην ξεπερνούν τα δύο λεπτά, λέει ο πρόεδρος, η κυρία Νούη. Για το πρώτο σημείο σας, πράγματι απαιτείται περαιτέρω σταθεροποίηση του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού πρέπει να τον κάνουμε ακόμα πιο ισχυρό. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Έχουμε 19 διαφορετικούς εθνικούς τραπεζικούς τομείς σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές τις εποπτικές και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο για, τις, την αναδιοργάνωση της αγοράς, της τα κτλ. Κάτι το οποίο απαιτείται στην Ευρώπη γιατί είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πάρα πολλές τράπεζες, πάρα πολύ μεγάλη προσφορά πιστοτικών υπηρεσιών και θα πρέπει να υπάρξουν συγχωνεύσεις και θα πρέπει να είναι και διασυνοριακές δεν είναι ρόλος των εποπτικών αρχών να λένε ποιες οι συγχωνεύσεις είναι καλές και ποιες δεν είναι καλές. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Οι επενδυτές και οι συμμετέχοντες, οι εμπλεκόμενοι στις αγορές είναι αυτοί οι οποίοι θα κρίνουν και θα αξιολογήσουν. Στα πλαίσια του ενιαίου μηχανισμού όμως εμείς θέλουμε να δράσουμε όσο μπορούμε καλύτερα έτσι ώστε να μην υπάρχουν και να προλαμβάνουμε τα εμπόδια στις συγχωνεύσεις αυτές τις διαμεθοριακές πιέζουμε περαιτέρω για ακόμα περισσότερες τέτοιες μορφές συγχώνευσης στο μέλλον. Κινούμεθα, κινούμεθα αργά, αλλά κινούμεθα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε οι εποπτικές δράσεις και ο ρόλος των εποπτικών αρχών θα βοηθήσουν αυτήν την βελτίωση της δομής του πιστοτικού συστήματος, της αύξησης της ρευστότητα, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο. Είδαμε γενικότερα την Ευρώπη και την Ευρωζώνη να βελτιώνεται στον τομέα αυτό. Σχετικά με το έντις. Κοιτάξτε, κινείται τουλάχιστον, το συζητάμε ακόμα μείωση των κινδύνων θα πρέπει να γίνει αναγνωρίζοντας παράλληλα την αύξηση της έννοιας της αρχής της αλληλεγγύης. Ήδη παρέχουμε ε, μέσω του SRM και του SSM ε, αρκετά στοιχεία μείωσης του κινδύνου. Το νομοθετικό πακέτο το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί τάχιστα, το TILAC, το NFRS, που θα πρέπει να ολοκληρωθούν τάχιστα. Ε, νομίζω ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορώ να είμαι πιο σαφής. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε μία φάση τώρα όπου όσο πιο γρήγορα μπορέσουμε να κινηθούμε ε, προς την ακόμα περισσότερη αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο το καλύτερο και νομίζω ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια βρίσκονται ακριβώς στη μέση αυτών των προσπαθειών και θα πρέπει να ε, εντείνουμε τις προσπάθειές μας αντίστοιχα. Για τα μη εξυπηρετούμενα χρειαζόμαστε χρόνο, μιλάμε για τις ροές ε, και όχι ε, τις, τα στόκ των μη εξυπηρετούμενων στην πρόταση προσθήκης εμείς μιλάμε για την ανάγκη μη δημιουργίας νέων, μη ακάλυπτων, ε, νέων ακάλυπτων ε, μορφών έκθεσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλωσορίζω και εγώ την ε, κυρία Νούη. Θα ήθελα να θέσω τρία ακόμα ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε. το πρώτο ε, αφορά ένα σκάνδαλο με υπονθήκες στην Ελλανδία όπου ε, διαπιστώθηκε ότι οι κύριες ελληνικές τράπεζες οι οποίες ε, περισσότερες από αυτές έχουν υποβληθεί σε εποπτεία έχουν ουσιαστικά συνεργάστηκαν μεταξύ τους προκειμένου να υφαρπάξουν ε, εκατομμύρια ουσιαστικά ε, από τα χρήματα που έχουν επενδύσει σε υποθήκε οι διάφοροι καταναλωτέ. Οπότε θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η αντίδραση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με αυτό το σκάνδαλο. Έχει αναλάβει κάποια δράση και έχει τι απαραίτητε εξουσίε για να λάβει αυτή τη δράση ε, προκειμένου να διαρευνήσει καλύτερα τι τις αυτών των τραπεζών οι οποίε είχαν υποβληθεί σε την εποπτεία. Δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω αφορά τα ε, μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ε, την προσωρινή πρόταση που κάνατε. Ε, συμφωνώ με κάποιες από τις κριτικές που ασκήθηκαν σε ό,τι αφορά την πρόταση του Επόπτου Οικονομικού Μηχανισμού σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ότι δηλαδή οι απαιτήσει που προβλέπονται εκεί σε αυτό το μηχανισμό δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις υφιστάμενες διαφορές μεταξύ των διαφορετικών κρατών μελών. Και επίσης το μηχανισμό SSM αναφέρεται στον κανονισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων για την ω βάση σε ό,τι αφορά την εκτίμηση των ε, εξυπηρετούμενων ε, δανείων. Ε, ωστόσο, για μένα το γεγονός ότι γίνεται μια προσπάθεια από EBD, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Επιτροπή για την αξιοποίηση των ε, νοσιακών κοντιλίων ε, για την αντιμετώπιση αυτών των ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων σημαίνει ότι θα έπρεπε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει περισσότερες εξουσίες, περισσότερο λόγο σε ό,τι αφορά αυτές τις αποφάσεις γιατί είναι κυρίως πολιτικού χαρακτήρα αυτές οι αποφάσεις και δεν είναι τεχνικού προκειμένου να λαμβάνονται σχετικέ αποφάσει από επόπτε και από άλλε ρυθμιστικές αρχές. Τέλος, όπως γνωρίζετε εσείς οι έφτασαν πρόσφατα σε μια ε, ε, ε, συμφωνία σε ό,τι αφορά την προσωρινή συμφωνία, σε ό,τι αφορά το συνολικό εναγωμένο κίνδυνο CRR και το σχετικό διεθνέ πρότυπο χρηματοοικονομική αναφορά 9 το FRS. Και έχει προβλεφθεί εκεί μια περίοδο 5 ετών. Οπότε θα ήθελα να ξέρω ποιος, ποια είναι η άποψη τη του σε σχέση με αυτή την προθεσμία των 5 ετών και τι ε, ε, ε, αυτό σημαίνει επακριβώς αν θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Ναι. Σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο με τις υποθήκες τράκερς στην ε, να εξηγήσω λίγο στους πολίτες το τι ακριβώς συμβαίνει. Στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής κρίσης, οι Ιρλανδικές τράπεζες παρήχαν δάνεια τα οποία παρακολουθούσαν ακριβώς τα ε, ε, επιτόκια της ε, Ευρωπαϊκής Θετικής Τράπεζας. Γι' αυτό ονομάστηκαν και τράτερ. Δηλαδή όταν μειώναν, μειώνονταν τα σχετικά επιτόκια καθίστονταν και τα σχετικά επιτόκια πολύ και εκείνα με τη σειρά τους σε κάποιες σημαίες γίνονταν αρνητικά πράγματα, το οποίο είχε βέβαια και πολύ δεν είχε καλό αντίκτυπο ε, στην, ε, στη φήμη τους. Δηλαδή χρησιμοποίησαν ουσιαστικά πρακτικές αυτές οι τράπεζες οι οποίες ε, βρίσκονταν εκτός των συμβατικών τους, των όσων είχαν συμφωνηθεί συμβατικά με τους επελατές τους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αρμόδια μόνο για το τμήμα του Prudential Supervision, για την εποπτεία, δηλαδή την Prudential. Τα υπόλοιπα αφορούν αρμοδιότητες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Ε, το γεγονός δηλαδή ότι ε, ε, κάποιοι δανειοληπτικοί οργανισμοί στο πλαίσιο αυτών των υποθηκών δεν σεβάστηκαν τα όσα προβλέπονταν συμβατικά με τους πελάτες τους είναι κάτι το οποίο αφορά τις εθνικές δεσμιστικές αρχές, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση την Εθνική Τράπεζα της Ιρλανδίας και όχι την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τώρα, είναι προφανές ότι όταν εμείς διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια τράπεζα η οποία ακριβώς ε, προβαίνει σε κάποιε παραβάσει, δηλαδή υπάρχουν ζητήματα εδώ σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών, προφανώ για του επόπτε, του potential επόπτε, ε, ε, προκύπτει ένα ζήτημα, αρχίζουν να παρακολουθούν καλύτερα τα ζητήματα δηλαδή συμμόρφωσης και δίνεται περισσότερη έμφαση σε αυτές τις πτυχές ελέγχου αυτών των τραπεζών. Δηλαδή υπάρχει αντίκτυπο σε ό,τι αφορά το Prudential Supervision από την πλευρά μα, αλλά δεν αποτελεί δική μας αρμοδιότητα η, μια τέτοια πρακτική από αυτέ τι τράπεζε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, λαμβάνω υπόψη μου ότι και εσείς συμμερίζεστε την κριτική που αστήθηκε και η, η Ιρλανδία και οι πρώτε τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, έχουν βρεθεί στην αιχμή του δόρατο αυτή τη προσπάθεια τη γνωρίζω πω ο έχει πράγματι κάνει πολύ καλή δουλειά ε, σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, οπότε θα πρέπει να βασιστούμε, βασιστούμε στις βέλτιστες, αν θέλετε, πρακτικές, στις πλέον επιτυχημένες πρακτικές σε ό,τι αφορά την εποπτεία σε, άλλες, σε άλλα κράτη-μέλη. Τώρα, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να μας βοηθήσει για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την έκθεση σε με εξυπηρετώμενα δάνεια, προφανώς είναι πολύ ευπρόσδεκτη η υποστήριξή του, γιατί αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σε ό,τι αφορά την ε, καθυστέρηση, την παράταση της εφαρμογής του ΑΕΦΑΡΕΣ 9, ε, ε, εγώ θα πρέπει να πω ότι συμμετέχω σε αυτές τις εργασίες εδώ και περισσότερο από 9 έτη και συνεργάζομαι από τις αρχές του 1991 με την Επιτροπή της Βασιλείας ως μέλος και πάντοτε ανέκαθεν θέλαμε να καλύπτονται ε, όχι μόνο οι ζημίες οι οποίες έχουν λάβει χώρα, incurred losses, αλλά και οι αναμενόμενες ζημίες, expected losses. Και αυτό βέβαια είναι ε, σημαντικό, γιατί ε, πάντοτε και οι σχετικοί υπολογισμοί για τις κεφαλαϊκές αποτέσεις γίνονται και σε σχέση με τα μελλοντικά, τα αναμενόμενα, τις αναμενόμενες ζημίες. Άρα, όταν λέμε ότι θέλουμε 10 συμπληρωματικά έτη από τη συμφωνία, προκειμένου να επιτύχουμε ένα πρότυπο σε ό,τι αφορά τους, και τις εποπτικές αρχές είναι αρκετό ο Προφανώ ε, Προφανώς ε, δεν συμφωνούμε όλοι σε όλα τα ζητήματα, αλλά σε ό,τι αφορά το τμήμα του Prudential, τουλάχιστον το αρχικό σοκ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο να τύχει διαχείριση. Ε, δεν προβλέπουμε δηλαδή από εκεί και μετά συμπληρωματικό phasing αλλά phasing in για το πρώτο σοκ, ναι, θεωρώ πω είναι μια σοφή προσέγγιση, ακόμα και αν εγώ προσωπικά βέβαια δεν θέλω να περιμένουμε πάρα πολύ. Ε, μάλιστα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτο σημείο, κυρία Νουή, θέλω να αναφερθώ στην ε, νομική ε, κρίση του Κοινοβουλίου πάνω στην πρόταση προσθήκης. Την πήρατε χθε και πρέπει πρώτα να την αξιολογήσετε, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ε, ποιες είναι οι συγκεκριμένες σας αρμοδιότητες, ποια είναι η εντολή σας, ιδιαίτερα σε ευαίσθητα θέματα όπως αυτά, απαιτείται να υπάρχει μια σαφής θεσμική κατανομή αρμοδιοτήτων και εσείς δεν θα πρέπει να ξεπεράσετε τις δικές σας. Μπορούμε να επανέλθουμε στο θέμα αυτό ιστερότερα και να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποιους κανόνες που δεν αφορούν μόνο τις εποπτικές αρχές Σχετικά τώρα με τα μη εξυπηρετούμενα. Νομίζω ότι η τάση ε, που υπάρχει να υπογραμμίζουμε ακόμα περισσότερο το θέμα αυτό επηρεάζει αρνητικά τις αγορές. Η αγορά των MPL τώρα βρίσκεται σε μια πολύ ευαίσθητη φάση γιατί προσπαθούν οι τράπεζες να διαχειριστούν αυτά τα προβληματικά στοιχεία και να αποφύγουν μεγάλες απώλειες και κάθε φορά που κυκλοφορούν ευαίσθητες πληροφορίες γύρω από τα θέματα αυτά πέφτουν οι τιμές των μετοχών και χειροτερεύει η κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια πιο υπεύθυνη συμπεριφορά σε σχέση με την κυκλοφορία των πληροφοριών αυτών. Οι τράπεζες υφίστανται όλο και μεγαλύτερες απαιτήσεις κεφαλαιοχικές εξακολουθούν να αναζητούν κεφάλαια και είδαμε τι έγινε με τα παράγωγα και τη γνωμοδότηση της ΕΣΜΑ στο τέλος Οκτωβρίου. Βρισκόμαστε σε μια αγορά 455 δις, ενώ τα NFL είναι γύρω στα 800 δις. Λοιπόν, δεν βλέπω να είμαστε συγκεκριμένοι απέναντι στα προβλήματα αυτά, τα οποία είναι μόνιμα και συστηματικά και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί αν πρέπει να βασιζόμαστε αποκλειστικά στα μη ρευστά στοιχεία, ρευστοποιημένα στοιχεία και από τον τομέα των παραγόγων, τότε οι τράπεζες που είναι εκτεθειμένες απέναντι στα θέματα αυτά θα μας κάνουν να πληρώσουμε ακριβά την κρίση. Και ε, θα πρέπει ακριβώς να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να κερδίσει από την ιστορία αυτή των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αυτούς οι οποίοι προσπαθούν με καταχρηστικό τρόπο να το εκμεταλλευτούν αντίθετα με αυτούς που θέλουν να το επιλύσουν. Σας ευχαριστώ. Ακούστε, ας ελπίσουμε ότι οι συζητήσεις, οι σημερινές διευκρίνησαν κάποια πράγματα. Ανατράπεζα γίνεται η ανάλυση. Το ξαναλέω και τα εποπτικά μέτρα ανατράπεζα. Ένα πιλωτικό εργαλείο. Βεβαίως ε, υπάρχουν κάποιοι, ε, κάποιοι θεσμοί ε, που θεωρούν ότι μοιάζει με τον ε, πρώτο πυλώνα, δεύτερο δεύτερος αυτό είπα πριν, δεύτερος πυλώνας, πυλαρτού. Κάποια στιγμή είπατε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες μπορούν να διαχειριστούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ε, αποφεύγοντας τις απώλειες. Ε, ενδέχεται όμως ορισμένες φορές να αντιμετωπίσουν απώλειες ε, στα πλαίσια των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ιδιαίτερα αν δεν είναι αρκετά καλυμμένες. Θα πρέπει να αποφασίσουν πότε και πώς ε, θα κάνουν αυτές τις εκαθαρίσεις ε, των τιμολογίων τους. Ε, αυτό είναι κάτι επίπονο, αλλά είναι απαραίτητο. Διαβάστε την ομιλία του Πρόεδρου της ΕΚΤ την Τρίτη που καθιστά σαφέ ότι τα στατιστικά στοιχεία τη ΕΚΤ που είναι εξαιρετική ποιότητα αποδεικνύουν ότι οι τράπεζε που είναι επιβαρημένε με μη εξυπηρετούμενα δάνεια τελικά δανείζουν λιγότερα στι επιχειρήσει και στι μικρομεσαίε επιχειρήσει τη Ευρωζώνη. Σε ό,τι αφορά τα, τα στοιχεία επίπεδου 3, όπω έχω πει πολλέ φορέ, εμεί εξετάζουμε όλου του τύπου κινδύνου από όπου και αν προέρχονται. Το κάνουμε αυτό πολύ προσεκτικά και πολύ σοβαρά και για τα περιουσιακά στοιχεία ε, επίπεδου 3. Εξετάζουμε τα μοντέλα τιμολόγησης, ε, τις πτυχές ε, κινδύνου για την αγορά, τακτικά το κάνουμε αυτό και κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης του ιστορικού μοντέλου αποτελεί μέρος και του ΣΡΕΠ e της διαδικασίας αναθεώρησης. Ε, έχουμε ένα αυξημένο αριθμό αποστολών, επιθεωρήσεων σε ό,τι αφορά τα στοιχεία επίπεδου 3. Ε, μετά την κρίση οι τράπεζες ε, ούτως ή άλλως έχουν λιγότερη όρεξη για τέτοιου είδους κινδύνους διότι κάηκαν αλλά άνθρωποι είμαστε και οι τραπεζίτες είναι άνθρωποι και νομίζω ότι σε κάποια φάση θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα θέματα αυτά και γι' αυτό ακριβώς κυκλοφορήσαμε ε, και κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την μοχλευμένη χρηματοδότηση έτσι ώστε να αποφύγουμε την λήψη περαιτέρω κίνδυνων και να σας πω παράλληλα ότι στα πλαίσια του ορισμού ε, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας σε δεύτερο επίπεδο και σε τρίτο επίπεδο σε σχέση ε, με τις κεφαλαιοχικές απαιτήσει έχουμε το complexity element και το resolvability element τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Αυτό ε, νομίζω θα μας αποτρέψει να αποτύχουν ε, και να περάσουν σε διαδικασία εξυγίανσης περισσότερες τράπεζες λόγω των κινδύνων των αγορών εφόσον δεν αντιμετωπιστούν τα MPL στο μέλλον. Μπερνάρ Μονό έχει το λόγο, παρακαλώ. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε. Εδώ και κάποιες εβδομάδες ε, ζητάτε μείωση του τραπεζικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέτε ότι είναι πολλές οι τράπεζες που δεν είναι αρκετά ε, δεν, έχουν αρκετά, δεν είναι αρκετά επικερδείς και έχουν και πολύ προσωπικό. Είπατε μάλιστα στη Μαδρίτη πριν μερικές ε, μέρες ότι πρέπει να εξαφανιστούν μια σειρά από χρηματοπιστωτικά όργανα ε, μέσω πτώχευση. Αυτό πραγματικά με εποπτική αρχή να εύχεται πτωχεύσει δεν το καταλαβαίνω. Λέτε στην Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει τι πτωχεύσει διότι έχει το μηχανισμό ε, ε, ενιαία εξυγίανση. Όμω δεν είναι πολύ μεγάλο ο κίνδυνο όταν οι χώρε είναι ήδη υπερχρεωμένε, δεν μπορούν να υποστηρίξουν τι τράπεζέ του. Υπάρχει ένα ενιαίο ταμείο εξυγίανση το οποίο είναι σχεδόν άδειο και τα MRL δεν υπάρχουν. Επίση, μα μιλάτε, συγκρίνετε την Αμερική και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν πρέπει να αντικαταστήσουμε την χρηματοδότηση των, από τι τράπεζε και να έχουμε περισσότερε χρηματαγορέ. Μια μέση, μέσω μεγέθου τράπεζα, τράπεζα σε τοπικό επίπεδο δεν μπορεί να αναλύσει καλύτερα σε το οικονομικό ε, ε, πλαίσιο από ότι ένα μακρινό ε, επενδυτή. Επίση, ζητάτε συγχωνεύσει των τραπεζών και ήδη δυνατόν διασυνοριακές συγχωνεύσεις. Το πρόβλημά μου εδώ είναι το ίδιο. Μια τοπική τράπεζα μπορεί, μπορεί πολύ καλύτερα να χρηματοδοτήσει μικρομεσαίε επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία από ότι ένα ε, πολυεθνικός γίγαντας που μόνο, το μόνο που θα θέλει να κάνει είναι να μειώσει το κόστο. Το να προωθήσουμε τι συγχωνεύσεις διασυνοριακέ θα έχει και άλλε αρνητικέ επιπτώσεις. Τελευταίο ερώτημά μου εδώ. Η Lehman Brothers ε, είχε ξεκίνησε την, τραπ, την, την κρίση του 2008 διότι είχε μία διασύνδεση στο τραπεζικό τομέα. Ε, θέλουμε πραγματικά να αυξήσουμε τη διασύνδεση τη διασυνοριακή στην Ευρώπη. Ποια είναι τα ωφέλη. Ε, πρέπει μόνο να ικανοποιήσουμε ε, ιδεολογικά ε, την εξάλληψη των συνόρων. Μήπως θα πρέπει ε, να έχουμε να, να μπορέσουμε να κατακαιρματίσουμε τους κίνδυνους όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό ανέφερε και το παγκόσμιο κριτήριο του ΣΥΦΗ ε, που ήταν κατά της διασύνδεσης αυτής. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου θέλετε τα ερωτήματα αυτά, διότι ε, ορισμένε φορέ μπορεί να μην καταλάβατε, να, να μην έγιναν κατανοητά αυτά που είπα εγώ στα αγγλικά στην Ισπανία τότε, διότι εγώ δεν είπα τέτοια πράγματα. Ε, θα συνεχίσω στα αγγλικά για τους υπόλοιπους. Είναι πραγματικά δύσκολες αποφάσεις αυτές. Είναι επίπονες για τους επενδυτές, για τους καταθέτες, για τις άλλες τράπεζες, διότι αυτό έχει και ε, διαχέεται ε, μια πτώχευση και πρέπει να αποφεύγουμε την πτώχευση των τραπεζών. Όμως, εμείς δεν έχουμε την εξουσία, δεν είναι δουλειά μας να προλάβουμε την κάθε πτώχευση τράπεζας. Είμαστε σε ένα περιβάλλον ελεύθερης αγοράς. Εάν μια τράπεζα εθελοτυφλή δεν ακούει τις εποπτικές αρχές, προτιμά ε, να παίρνει ε, τυχοδιοκτικές αποφάσεις ε, επενδυτικές, δεν πρόκειται ε, να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την πτώχευσή τους. Σε ό,τι αφορά την, ε, την ανάγκη ε, ενοποίησης και τις πολλές τράπεζες που υπάρχουν στην Ευρώπη, αυτό δεν ισχύει, δεν ισχύει για όλες τις χώρες βέβαια, στην Ευρώπη όμως συνολικά. Είναι αλήθεια, εάν το συγκρίνουμε με το ΑΕΠ της περιοχής, ε, της περιοχής αυτής, ε, δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση με άλλες χώρες ε, ή άλλες περιοχές. Ένας αριθμός ε, ευρωπαϊκών τραπεζών δεν, δεν κερδίζουν ποσά ανάλογα με το κεφάλαιό τους. είναι μη βιώσιμες μακροπρόθεσμα. Πρέπει λοιπόν να αξιολογηθεί η βιωσιμότητα του business model αυτών των ε, τραπεζών και αυτό δείχνει ότι υπάρχουν, υπάρχει, υπάρχει υπερβολική πρόσφορα τραπεζικών υπηρεσιών ε, και να παρθούν μέτρα γι' αυτό για να μην υπάρξουν πτωχεύσεις ακριβώς. Μπορεί να παρθούν μέτρα σε εθνικό επίπεδο βέβαια, δεν έχουμε καμιά αντίρρηση και να το λάβουν, λάβουν χώρα συγχωνεύσεις ε, σε εθνικό επίπεδο ε, μέσα σε μια χώρα. Είναι πιο εύκολο συνήθω, είναι πιο εύκολο να βρεθούν συνέργειε, ε, ε, δεν μπαίνουν και ζητήματα σχετικά με τη ρευστότητα κεφαλαίων. Ε, Όμω βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου είναι κρίμα οι τράπεζες να μην εκμεταλλευτούν ε, τις συνέργειες που υπάρχουν, ο συστημικός χαρακτήρας μπορεί πλέον να αξιολογηθεί ευρύτερα, στα πλαίσια της Ευρωζώνης, όχι μόνο αναχώρα. Ναι, λοιπόν, χρειαζόμαστε ενοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Ε, η αγορά θα αποφασίσει πώς θα γίνει αυτό. Η δουλειά των εποπτικών αρχών είναι να εξετάσουν αυτές τις συγχωνεύσεις έτσι ώστε να είναι βέβαιες ότι είναι υγιείς, ότι είναι σταθερές, ότι είναι ασφαλείς και θα προσκομίσουν ωφέλη στους καταθέτες και στους επενδυτές. Ε, δεν πρόκειται εμείς όμως να πούμε ε, πώς θα γίνουν οι συγχωνεύσεις. Ε, καλύτερα όμως να έχουμε συγχωνεύσεις παρά να εθελοτυφλούν οι τράπεζες και να πτωχεύουν. Ο κ. Κίτσος έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Νουή για την ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση. Θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σας ε, για την εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού τομέα, διότι στην Ελλάδα έχει σημειωθεί πρόοδος ε, σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική κατάσταση, όμως η κατάσταση στον τραπεζικό τομέα, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, ε, παραμένει αρκετά εύθραυστη υπάρχουν μεγάλε αμφιβολίε ό,τι αφορά το κατά πόσο το, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να αντιμετωπίσει το, το υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση διστάζει να, δίστασε να εφαρμόσει την συμφωνημένη πολιτική που προβλέπει ε, τις εξώσεις ε, και τις, ε, κατασχέσεις τραπεζών διότι δεν μπορεί να το κάνει διότι άλλα υποσχέθηκε στο ακροατήριο το πολιτικό του. Ε, επίσης θα περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να, μπορέσει, να μπορέσουν οι τράπεζες ε, να επενδύσουν την οικονομική ανάπτυξη, στην οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Για άλλη μια φορά ε, θα, δεν θα έχουμε αρκετό χρόνο για να προχωρήσουμε στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τα νέα εξυπηρετούμενα δάνεια και, και τα παλαιά, ε, έχει δημιουργηθεί ένα άγχος, ένα στρες ε, στην, στο τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης και αυτό έχει συνεισφέρει στην μείωση, την περαιτέρω μείωση της τάξης του 25 με 30% των αξιών της στο χρημα, των μετοχών στο χρηματιστήριο. Φτάνουμε, πλησιάζουμε σε ένα σημείο όπου οι αρμόδιες τραπεζικές αρχές οι ευρωπαϊκές θα πρέπει να βρουν ε, δημιουργικούς τρόπους για να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση και τη βελτίωση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα. Ποια είναι η αποψία σας επ' αυτού. Θα πρέπει να δεχτούμε ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς ή θα πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες με συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσουμε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και να μην υπάρξουν περαιτέρω επιπλοκές. Ευχαριστώ πολύ. Ακούστε, οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη κάνει σημαντικές προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Βεβαίως λόγω του μεγέθους ε, του προβλήματος είναι δύσκολο. Επίσης ε, χρειάστηκε να αλλάξει το νομικό πλαίσιο ε, για να μπορέσει πιο σοβαρά να αντιμετωπίσει το ζήτημα, ε, το σύστημα. Αυτά όμως έχουν γίνει τώρα και ήρθε η ώρα να δρέψουμε τα ωφέλη από αυτές τις αλλαγές και να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης να σας θυμίσω ότι οι ελληνικές τράπεζες όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, τράπεζες της Ευρωζώνης ε, ελέγχουν, θα ελεγχθούν μάλλον από, το, από την EBA το 2018. Θα υπάρξει stress test και θα αξιολογηθεί η κατάσταση για τις τράπεζες αυτές και για τις υπόλοιπες. Και έτσι θα γνωρίζουμε και καλύτερα κατά πόσο οι προσπάθειες έχουν αποφέρει καρπούς και τι μένει να γίνει. Να πω επίσης ότι βεβαίως δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες στην αντιμετώπιση των προβλημάτων σε διάφορες χώρες. Πάντα κάποιες τράπεζες ε, κινούνται πιο γρήγορα. Αυτό ισχύει και στην Ελλάδα. Τώρα, κατά πόσο πρέπει να συνεχίσουμε, ε, κατά πόσο τα πράγματα βαίνουν ομαλά στην Ελλάδα, όχι, δεν μπορεί να το πει κανεί αυτό. Αλλά αυτό, δεν αφορά, αυτό αφορά όμω και την Ευρωζώνη γενικότερα. Έχουμε μια σειρά προκλήσει να αντιμετωπίσουμε. Βεβαίω υπάρχει το θέμα τη έκθεση στα μη εξυπηρετούμενα δανεία, αλλά υπάρχει και το θέμα του κέρδου των τραπεζών. Πρέπει να μπορέσουν να είναι επικερδεί τράπεζε, όπω είπα νωρίτερα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Όχι. Ωραία. Ο κ. Σίλβα Περέιρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σωστά υπογραμμίσατε ότι οι προτάσεις σας για τα NPL είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει πάρει την τελική μορφή, μπορεί να βελτιωθεί και να λάβετε υπόψη σας παρακαλώ σοβαρά τα αποτελέσματα της ε, διαβούλευσης. Νομίζω ότι ε, χρήζει περαιτέρω βελτίωση η πρότασή σας και νομίζω ότι το αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης θα είναι μια διαφορετική πρόταση, πιο εξισορροπημένη, η οποία θα πρέπει εκ νέου να τεθεί σε διαβούλευση βέβαια. Νομίζω ότι αυτά τα οποία προβλέπει η πρότασή σας είναι λανθασμένα, δημιουργούν μια μόνιμη θεσμική αστάθεια. Είναι αντιπαραγωγικές οι προτάσεις σας και σε σχέση με τα NPL και θα έχει πάρα πολλές αρνητικές επιπτώσεις στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην οικονομική ανάκαμψη. Έχω τρία βασικά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση επιπτώσεων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ομολογώ με εκπλήσει. Εσείς κάνετε μια θεσμική δήλωση για την επάρκεια την κεφαλαιουχική και σε επίπεδο ενεργών του τραπεζικού τομέα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη βέβαια σημασία. Οι συνέπειες αυτών των προτάσεων θα είναι η πώληση ε, στοιχείων ιδιόκτητων που θα οδηγήσει σε πολλά προβλήματα και στους ισολογισμούς των τραπεζών, θα δημιουργήσει μια πιθανότατα αύξηση των μη εξυπηρετούμενων, οι νέες απαιτήσει θα επηρεάσουν αρνητικά την δανειοληπτική δυνατότητα των τραπεζών και θα δημιουργηθεί ένας περαιτέρω συστημικός κίνδυνος που θα οδηγήσει στην αστάθεια τη δημοσιονομική ε, και όλα αυτά χωρίς αξιολόγηση επιπτώσεων. Τώρα δεύτερον, οι μη δεσμευτικές σας προτάσεις. Ε, δεν νομίζω ότι είστε ιδιαίτερα πιστικοί εδώ. Φυσικά και είναι δεσμευτικοί. Ε, μια ποσοτική προοπτική είναι ουσιαστικά ένας κανόνας. Ο μηχανισμός ο οποίος προβλέπεται επιβεβαιεί τον δεσμευτικό χαρακτήρα του κανόνα αυτού και εσείς ε, ε, προβλέπετε ε, κάποια νέα οπτικά μέτρα τα οποία επιβεβαιώνουν το δεσμευτικό χαρακτήρα της πρότασης. Όταν εμείς ελέγχουμε την συμβατότητα της πρότασης με τους ισχύοντες κανόνες, αυτό το κάνουμε κατά περίπτωση και αυτό μπορεί να δημιουργήσει ενδιάμεσα προβλήματα. Έχουμε να κάνουμε με μία πρόταση η οποία είναι αρνητική και δεσμευτική δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα απαιτούμενα επίπεδα επάρκειας, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση, οπότε συνολικά αυτό θα είναι αρνητικό. Και θα έχει και αναδρομική θα έλεγα δράση αντίθετα από αυτά που είπε ο κ. Κωνστάνθιο, αυτά θα εφαρμοστούν και στα ισχύοντα δάνεια και όχι μόνο στα νέα δάνεια. Ε, θα ασχοληθούν λοιπόν και με το σύνολο των δανείων τα οποία θα ταξινομηθούν στο μέλλον όσο μη εξυπηρετούμενα και αυτό θα δημιουργήσει αναδρομικά πάρα πολλά προβλήματα και έχουμε πρόβλημα και διαδικαστικό με την θέση σε ισχύ, αλλά ο αναδρομικός χαρακτήρας είναι το πιο προβληματικό στοιχείο της πρότασής σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήσατε λέγοντας ότι η διαβούλευση είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ε, αυτό κάνουμε, προφανώς και το κάνουμε αυτό συστηματικά και φυσικά όλα τα σχόλια τα οποία θα λάβουμε θα τα λάβουμε σοβαρά υπόψη. Τώρα δεν έχει υπάρξει μελέτη επιπτώσεων. Κοιτάξτε, μιλάμε για τα νέα NPL, τα νέα μη εξυπηρετούμενα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν υπάρχουν ακόμα. Δεν μιλάμε για το στόκ των υπαρχόντων δανείων. Εκεί θα μπορούσαμε να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι επιπτώσεις. Αλλά εδώ είναι δύσκολο να τις αξιολογήσουμε. Μιλάμε για νέα NPL τα οποία θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια θετικά εξελισσόμενων οικονομικών συγκύριων και αυτό είναι πολύ περίπλοκο να το κάνουμε. Είπατε επίσης ότι η πώληση ιδιοκτητικών στοιχείων ε, προφανώς ε, ε, οι πωλήσει δεν θα δημιουργήσουν, αντίθετα θα ενισχύσουν τους ισολογισμούς των τραπεζών. Μιλάμε για δάνεια τα οποία είναι σε μια πρώτη φάση εντελώς ε, κερδοφόρα. Είπατε ότι δεν είμαστε πιστικοί όταν σας λέγουμε ότι δεν είναι δεσμευτικός ο χαρακτήρας των προτάσεών μας. Κοιτάξτε, θα προσπαθήσω και μέσω της διαβούλευσης να σας πείσω για τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα. Τι άλλο θέλετε να κάνω. Σας ευχαριστώ, Χούμπνερ. Ευχαριστώ. Δύο σύντομες ερωτήσεις σε σχέση με την αναθεώρηση του SSM. Ε, αυτή η έκθεση αναθεώρησης της Επιτροπής του Οκτωβρίου ε, σε γενικές γραμμές είναι θετική, εξαιρετικά θετική, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα που αναφέρει και κάποιες συστάσεις που κάνει. Οπότε θα ήθελα να σας θέσω σχετικά δύο ερωτήματα. Ε, σε αυτή την έκθεση η Επιτροπή λοιπόν σημειώνει ότι τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συχνά προβαίνει σε, μια σειρά από ταξινομήσεις ε, των εποπτευόμενων αυτών ε, ε, φορέων για μια σειρά από λόγους και η Επιτροπή θεωρεί πως θα είχε νόημα να είναι πιο διαφανής η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αυτήν την ταξινόμηση. Και επίσης αναφέρει ότι αυτή η διαφάνεια θα πρέπει να είναι πιο σαφής ειδικότερα σε ό,τι αφορά ε, τις αποφάσεις, σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση αφενός ε, και το, τι, ποια συνέχεια δίνεται ε, ακριβώς στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής με βάση αυτή την ταξινόμηση. Οπότε θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω τι έχετε σκεφτεί σχετικά, ποιε είναι οι δυνητικέ λύσει. Δεύτερο ερώτημα και πάλι σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του SSM είναι οι διαδικασίε που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο του εποπτικού μηχανισμού σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με το ΕΜΠΑ. Ε, υπάρχουν δηλαδή κάποιες συστάσεις ε, ε, προκειμένου να βελτιωθεί η συνοχή, να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις σε ό,τι αφορά τα ζητήματα συντονισμού και οπότε το ερώτημά μου σε σχέση με αυτό το ζήτημα είναι θεωρείτε πως πράγματι θα πρέπει να δώσετε μια συνέχεια σε αυτές τις συστάσεις της Επιτροπής ε, και τι ακριβώς έχετε σκεφτεί. Ένα ακόμα ερώτημα που δεν σχετίζεται άμεσα με την αναθεώρηση του SSM αλλά μάλλον σχετίζεται περισσότερο με την αντίκτυπο του Brexit και τα όσα θα συμβούν μέχρι τότε, είναι οι ε, επιχειρήσει επενδύσεων ε, κατοφυλάκιων, δηλαδή ε, investment firms. Γιατί τέτοιου είδου επιχειρήσεις μπορούν να, θα μπορούν να προσφέρουν ε, μία σειρά από υπηρεσίε ε, και κατά συνέπεια ενδέχεται να εμπίπτουν στι ε, διατάξει του κανονισμού σε ό,τι αφορά τι τεχνολογικέ απαιτήσει. Γνωρίζουμε πω η Επιτροπή έχει ξεκινήσει τις εργασίες τη σε ό,τι αφορά αυτέ τι επιχειρήσει χαρτοφυλακή. Οπότε ε, θα θέλαμε να ξέρουμε, εσεί συνεργάζεστε με την Επιτροπή, βρίσκεστε σε επαφή προκειμένου να αναγνωρίσετε κινδύνου σε ό,τι αφορά αυτέ τι επιχειρήσει στο δικό σα τομέα αρμοδιότητα. Ε, κυρία Σα ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση και την ανάγκη για περισσότερε διαφάνειε σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση που κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να σας καταδείξουμε ποια είναι η ταξινόμηση που χρησιμοποιούμε, αλλά θα ε, πρέπει να κινηθούμε βήμα προς βήμα και βρισκόμαστε ακόμα σε φάση προσεκτική. Ε, ανάλυσης προσωπική εξέτασης όλων των τραπεζών για να ξέρουν όλες οι τράπεζες που ακριβώς βρίσκονται στο πλαίσιο της αξιολόγηση και της ταξινόμησης ε, που γίνεται. Πάντοτε στο πλαίσιο της εποπτικής μας αρμοδιότητας. Μετά, ε, σε ό,τι αφορά την δημοσιοποίηση της μεθόδου ταξινόμησης, καταρχήν υπάρχει μια ε, συμφωνία εμπιστευτικότητα ε, μεταξύ των θεσμικών οργάνων, η οποία μα υποχρεώνει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ω προ τα στοιχεία που δημοσιοποιούμε. Και από εκεί και μετά, βέβαια, δεν μπορεί η εποπτική αρχή να τεθεί, αν θέλετε, δημοσίω σε κάποιο είδου ελέγχο. Οπότε πράγματι θα πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία εδώ. Πάντω το ελάχιστο το οποίο έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμή είναι το να γνωρίζει κάθε ε, τράπεζα σε ποια κατηγορία αυτή τη ταξινόμηση έχει περιληφθεί. Και πάντοτε ε, λέμε στις τράπεζες, εάν έχετε ερωτήσεις μπορείτε να θέσετε ερωτήματα, εάν δεν είστε ικανοποιημένοι ε, ε μπορείτε να θέσετε ερωτήματα στην EGD, και αν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντηση που θα λάβετε μπορείτε να απευθυνθείτε και σε μένα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά το ΕΜΠΑ και τη σχέση προφανώς ε, χαιρετίζω εδώ το, ε, το έργο που έχει κάνει σε ό,τι αφορά την, ε, τη ενιαία καθοδήγηση, σε ό,τι αφορά τους ενιαίους δηλαδή κανόνες. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει καθοδήγηση ΕΜΠΑ. Και έτσι εκ των πραγμάτων καλούμαστε να λάβουμε μία απόφαση για 19 κράτη-μέλη. Αναγκαζόμαστε, αν θέλετε, να αναλάβουμε τον ηγετικό ρόλο για το σύνολο της Ευρώπης. Δεν είναι ότι αυτό ισχύει ότι αυτό καλούμαστε να κάνουμε, ε, αλλά δεν μπορούμε να ζητούμε από το ΕΜΠΑ να ε, έχει καθοδήγηση για όλα τα επιμέρους ζητήματα. Οπότε, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου να υπάρχει μια ασυνέχεια, αν θέλετε, μεταξύ των εργασιών μας και αυτών του ΕΜΠΑ, είναι ε, πάντοτε να υπάρχει αλληλεγμένος. Για παράδειγμα, αν ασχολούμαστε πρώτοι με ένα ζήτημα, ε, τότε πάντοτε εξετάζουμε αν έχει κάνει ήδη ε, ο ΕΜΠΑ. Και αν πράγματι έχει γίνει κάτι από την πλευρά του ΕΜΠΑ, τότε εμεί δεν κάνουμε κάτι άλλο. Ακολουθούμε τα όσα έχει προβλέψει ο ΕΜΠΑ, γιατί προφανώ πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό ε, φορέα, οπότε προφανώ θα ακολουθήσουμε τα όσα προτείνουν. Αλλά έχουμε βέβαια μια κατάσταση τύπου πολλώνα 1, πυλώνα 2. Δηλαδή, αν έχουμε πολιτικέ οι οποίε εφαρμόζονται σε 19 κράτη-μέλη, τότε ε, δείχνουμε, δείχνει να αναδύεται αν θέλετε ένας ευρωπαϊκός τρόπος που κάνουμε τα πράγματα το ε, οποίο να, μην ε, συμβαδίζει να μην είναι ίδιος με αυτό που προτείνω εγώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου τις investment firms από το Ηνωμένο Βασίλειο, με βάση τους κανόνες επενδύσεων ε, προβλέπεται δυνατότητα για τα PRA να προβαίνουν σε εποπτεία τουλάχιστον ε, ως τραπεζικά ιδρύματα των, τουλάχιστον των μεγάλων ε, τέτοιων επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου. Υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα εποπτείας τους ω τραπεζικού ιδρύματο. δεν χρειάστηκε όμω να εφαρμόσουμε αυτού τους κανόνες μέχρι στιγμή, γιατί μέχρι στιγμή στο Λονδίνο έδρευαν όλε αυτέ οι μεγάλε επιχειρήσει ε, χαρτοφυλακίου από τι ΗΠΑ, από την Ασία ναι, ήταν πολύ μικρότερε οι σχετικέ επιχειρήσει ε, δηλαδή σε άλλε χώρε ή ήταν θηγατρικέ αυτών των αμερικανικών ευρωπαϊκών ε, ομιλών. Οπότε αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη φάση δύο προβλήματα. Εάν δεν υπάρξει αλλαγή στον κανονισμό που να προβλέπει ότι συστημικές επιχειρήσεις και βέβαια ο νομοθέτης αποφασίζει τι ακριβώς είναι συστημικό, ε, εάν δεν θα προβλέπεται λοιπόν η υποπτία αυτών των συστημικών επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου τραπεζικών ιδρυμάτων, θα υπάρξει ένα κενό ε, στην νομοθεσία. Και από εκεί και μετά βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος καταγερματισμού. Γιατί είχαμε εποπτεία σε επίπεδο PRL και ξαφνικά θα έχουμε τώρα 19 διαφορετικές εποπτικέ αρχές των κρατών μελών που θα εποπτεύουν ε, κάθε μία ξεχωριστά αυτέ τι επιχειρήσει. Και βέβαια ενδεχομένω κάθε μία από αυτέ τι εποπτικέ επιχειρήσει να μην έχει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη, την απαραίτητη εμπειρία ε, για την ε, ε, εποπτεία αυτών των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Ευχαριστώ κυρία Νούη. Έχω δύο ερωτήματα για σας. Πρώτα για το spread μεταξύ δύο μορφών ε, χρέους. Είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο σε ορισμένε περιπτώσεις. Αυτό το spread, αυτή η απόκληση. Το έχει εξετάσει το θέμα η εποπτική αρχή. Είναι πολύ υψηλή, υψηλό το επίπεδο κινδύνου στην συνολόγο τράπεζες ή μπορεί να είναι αποτέλεσμα ε, σε ε, το υπρόεδρεσμα κάποιων όρων που απλά μπλέκουν τα πράγματα και τα θολώνουν ε, και είναι θέμα ονομασίας δηλαδή και μπορεί κάποιοι να ετοιμάζονται να χτυπηθούν και να, από εκεί που περιμένουν. Το δεύτερο, CCP Oversight. Όπως ξέρετε εξετάζουμε την ε, εποπτεία των CCP που συνδέονται με την σταθερότητα των παγκοσμίων τραπεζών. Ε, ε η εποπτεία της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας της Μάλτας ε, είναι ευρωπαϊκή, ε, είναι όμως εφικτό να ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Στα πλαίσια του Brexit δεν πρέπει αυτά τα πράγματα να τα βελτιώσουμε στα πλαίσια του νομοθετικού κύκλου και να έχουμε μια ενιαία εποπτεία και μια ενιαία εξυγίωνση για τα CCPs. είναι μια διαδικασία που θα, απόφασεις που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή για το ποιο είναι το κατάλληλο ποσό. Ε, αυτή είναι η απόφαση που παίρνει κάθε τράπεζα ξεχωριστά. Συμφωνώ πάντως μαζί σας απολύτως ότι θα πρέπει να δώσουμε ασφάλεια στους επενδυτές. Όντως υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ διαφόρων κατηγοριών ε, προϊόντων ε, που δημιουργεί σύγχυση. Ε, και ο κανονισμός του, της BRD είναι απαραίτητο διότι έχουμε οδηγία ω τώρα και αυτό οδηγεί σε μεταφορά της οδηγίας με 19 διαφορετικού τρόπους και αυτό έχει ένα κόστος διότι ο επενδυτή πάντα υποπτεύεται ότι το πιο επικίνδυνο σύστημα είναι το ευρωπαϊκό. Και αυτό είναι που θα έχει αρνητικές, αυτό είναι ο λόγος αν κάτι δεν πάει καλά. Ε, θα πρέπει να, δώσουμε, να παρέχουμε όμως ασφάλεια στους επενδυτές, να, να γνωρίζουν ε, τι ε, είναι ασφαλές, τι δεν είναι, ε, μέσα στα διάφορα επενδυτικά προϊόντα. Να πω επίσης ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα για να, για να εξασφαλίσουμε ότι οι λιανοπολιτές πρέπει να καταλάβουν οι τι προστατεύει και τι όχι. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ένας λιανοπολιτής βάζει τις αποτελεσματικές μια ζωή σε μία μόνο τράπεζα χωρίς ε, ε, να είμαστε βέβαιοι αν αυτά τα χρήματα είναι ασφαλή σε ό,τι αφορά τώρα τις, το CCP και τον έλεγχό τους. Όντως ε, πρόκειται για συστημικές ε, συστηματικούς οργανισμούς, συστημικούς οργανισμούς είναι πολλές περίπλοκες επιχειρήσεις που έχουν πάει προς τα CCP, τα έχουμε στείλει εκεί, ε, δεν είναι αυτοκριτική βέβαια. Ε, εγώ προσωπικά, προσωπικά, όχι το SSM, δεν το έχει το SSM, πιστεύω ότι ο αμερικανικός τρόπος όταν ένα CCP δηλαδή είναι συστημικό ε, εποπτεύεται από τη Φέντο όπως μια συστημική τράπεζα είναι ένας πιο απλός τρόπος. Και η, η απλότητα συχνά οδηγεί στην αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την εποπτεία. Αυτή τη στιγμή όμως είναι πολύ οι εμπλεκόμενοι στα πλαίσια του ΕΜΙΡ. Και αυτό περιπλέκει τα πράγματα. Δεν έχουμε ε, συμμετοχή σε αυτές τις συναντήσεις ε, ε, ίσως επειδή έχει πολύ κόσμο ήδη ε, εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα χρειάζεται μεγαλύτερη χρειάζεται περισσότερη απλότητα παραδείγματος χάρη η δυνατότητα η ΕΣΜΑ να είναι υποπτική αρχή αυτά της CCP θα ήταν μια καλή λύση θα πρότεινα πάντως ε, να είναι όσο γίνεται πιο απλή διαδικασία, να μην είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν λόγο για αυτές τις λεπτές περιπτώσεις όταν πρέπει να δράσουμε σχετικά γρήγορα. Αυτή είναι προσωπική άποψη όμως. Ε, δεν έχει συζητηθεί το θέμα στα πλαίσια του SSM και του ε, Νικητικού του Συμβουλίου. Φούλβιο Μαρτουτσέλο έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η γνωμοδότηση που σας δόθηκε άλλωστε χτες καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πρόταση προσθήκης καθορίζει ένα μηχανισμό επί τη βάση του οποίου ένα, ένα όργανο υποχρεούται να υπακούσει στα επίπεδα τα οποία προβλέπονται από την ίδια προσθήκη η θα έλεγα παραβίαση ή μη τήρηση αυτών των επιπέδων θα κρυθεί σαν κάτι το αρνητικό στα πλαίσια των ελέγχων και της εποπτείας. Οπότε ουσιαστικά ο μηχανισμός είναι ουσιαστικά δεσμευτικός. Γιατί εσείς μας λέτε ότι ακριβώς αυτό το προσχέδιο προσθήκης δεν είναι δεσμευτικό, δεν το καταλαβαίνω. Και τώρα σε σχέση με το περιεχόμενο του αντέντουμ αυτού, η Επιτροπή Εποπτείας έχει κάνει μια αξιολόγηση των επιπτώσεων των ποσοτικών αυτών προσδοκιών όπως προβλέπονται μέσα στην προσθήκη. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό τότε γιατί αυτή η αξιολόγηση δεν τίθεται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως αυτό προβλέπεται από τη διοργανική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ε, το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η υποχρέωση κάλυψης πλήρως των μη εξυπηρετούμενων μετά από δύο χρόνια είναι ένας κανόνας πάρα πολύ αυστηρός. Ποια είναι η λογική η οποία ακολουθήθηκε για να πάρετε τη συγκεκριμένη απόφαση. Τώρα τα επτά χρόνια επίσης ε, για τα εγγυημένα καλυμμένα δάνεια είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να κάνει δεκτό, ε, ιδιαίτερα σε επίπεδο αναλογικότητας. Είδαμε χτες στο τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας όλες οι Ιταλικές τράπεζες οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο των τραπεζών που ασχολούνται με τα NPL είδαν ότι υπήρχαν, ε, ε, ε, σταμάτησε η διαπραγμάτευσή τους των μετοχών τους ενώ διότι η πτώση ήταν πάρα πολύ ταχύτατη ήταν ουσιαστικά και αυτό είναι καρπός της ανακοίνωσης την οποία κάνατε σχετικά με την προσθήκη. Λοιπόν, εσείς είπατε ότι το έγγραφε αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί μετά από όλες τις αξιολογήσεις. Μήπως αυτή η προσθήκη τελικά παίζει κάποιο ρόλο θα έλεγα παραποίησης της εικόνας της ε, πιστοτικής αγοράς σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι πράγματι, και το είπα ήδη, όλες οι, όλα τα θετικά σχόλια τα οποία θα λάβουμε θα τα λάβουμε πραγματικά υπόψη έτσι ώστε ε, να υπάρξουν τελικά ε, και από πλευρά κοινοβουλίου σαφείς νομικέ ρυθμίσει, για προτάσει για σαφεί νομικές ρυθμίσει. Δεν έχω μελετήσει το χθεσινό σα έγγραφο ακόμα, θα το κάνω. Τώρα γιατί ε, πήραμε τις αποφάσεις αυτές. Για τη διετή περίοδο είναι 180 μέρες στις Ηνωμένε Πολιτείες καταρχάς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να κατηγορηθούμε όσο πλέον ακραίοι στον κόσμο. Σχετικά με την επταετή περίοδο για τα καλυμμένα. Νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλη περίοδος για την συλλογή των εγγύσεων. Βλέπουμε ότι μερικές φορές τα νομικά, τα αρχικά κείμενα χάνονται. Κάτι το οποίο δημιουργεί μια κάποια αβεβαιότητα για την ανάκτηση των, των στοιχείων και μιας και η αβεβαιότητα αυτή αυξάνεται και το τίμημα ε, για ε, την απόφαση της τράπεζας προς πώληση των μη εξυπηρετούμενων καθίσταται λιγότερο ελκυστική. Συνεπώς οι δυσκολίες που έχουμε Ε, δείχνουν ότι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι τράπεζες δεν πρόκειται να εξαφανιστούν από τη μία, πλευρά στην, από τη μία στιγμή στην άλλη και τα μικρά προβλήματα τείνουν μετά από καθυστερήσεις χρονικές να μεγενθύνονται. Τώρα το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστούν σε εύθετο χρόνο. Ποιος είναι ο εύθετος χρόνος. Είναι θέμα αξιολόγησης και θα αρκεστώ στις προτάσεις σας για να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. έχω και εγώ κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα, εγώ καλωσορίζω την πρόθεσή σας που εκφράσατε εδώ ε, να μας ακούσετε και να αναγνωρίσετε ότι οι αλλαγές και οι βελτιώσεις είναι απαραίτητες ε, για να αποφύγουμε τη σύγχυση μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα και για να έχουμε μια πράγμα, ένα μηχανισμό που να αφορά την κάθε τράπεζα ξεχωριστά και να μην γίνεται αυτοματοποιημένα για όλες. Και εσείς αναγνωρίσατε ότι ο, ο μηχανισμός ε, συμμόρφωσης και εξήγηση ε, δεν φαίνεται να είναι ο κατάλληλος και θα πρέπει να αλλάχθεί. Χρειάζεται πραγματικά ε, προσέγγιση ανατράπεζα και για άλλους λόγους, διότι έγινε αναφορά στην αβεβαιότητα στην αγορά. Πρέπει να αποφύγουμε το μείγμα αυστηρών ε, απαιτήσεων και, και τη σύγχυση του πώς θα εφαρμοστεί αυτό, ε, αυτό το μείγμα μπορεί να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Διότι πρέπει να καθαρίσουμε και ε, τα λογιστικά στοιχεία και αυτό είναι πάντα επίπονο, αλλά ένα πράγμα είναι οι απώλειες που πρέπει βεβαίω να ελαχιστοποιηθούν και άλλο πράγμα είναι η μη αναγκαία ε, μείωση της αξίας. Ε, όλοι να γνωρίζουν ότι ε, τα, υπάρχουν, τα υπάρχοντα συστήματα δεν είναι τέλεια. Ο, ο αγοραστής ε, επικρατεί του πολιτή, ε, δεν είναι μηδενική λοιπόν η αξία. Εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα που θα, όπου θα μπορούσε να βοηθήσει μια προσέγγιση ένα τράπεζα. Η έκθεση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι μια κατηγορία ε, που έχει να κάνει με το παρελθόν με αυτά που, που, που τα ωφέλη υπάρχουν από παρελθόν και αυτά που δεν ενδέχεται να μην πληρωθούν δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ε, θεωρείται non-performing exposure, ας πούμε, αυτή η απώλεια. Και αυτό πρέπει να εξεταστεί. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες δανείων. Ε, και στην ασφαλή και στη μη ασφαλή διάστασή τους. Ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό. Και επίσης θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα σε αφορά τη διάδραση με τις λογιστικές αρχές. Ε, γνωρίζουμε πόσο ε, ε, απαιτητικό είναι το IFIS 9 και πόσο ε, φιλόδοξο. Όλοι θέλουν πέντε χρόνια μεταβατική περίοδο. Ε, τώρα λέμε ότι ένα περιουσιακό στοιχείο κατηγορίας 3 ε, στα πλαίσια του FS9 θα πρέπει να αξιολογείται ε, με βάση το προσδοκόμενο cash flow. Ε, εδώ ήδη κάνουμε κάτι χωρίς μεταβατική περίοδο που πάει πέρα από, τις λογιστικές αρχή, από μια λογιστική αρχή που ήδη είναι πολύ αυστηρή και που θέλει πενταετή περίοδο μετάβασης. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε. Δεν πρέπει εδώ να αποτρέψουμε ε, την ε, ενοποίηση των τραπεζών, αλλά θα πρέπει να είναι σαφής, σαφής διαχωρισμός μεταξύ της ευθύνης των πολιτικών αρχών και των πολιτικών ε, των βιομηχανικών. Είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι Σοβιετική Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν η αγορά ε, να κάνει τη δουλειά της. Ε, εφαρμόσουν βεβαίως οι επόπτες τα, τους κανόνες, να έχουν τις προτιμήσεις τους, αλλά από εκεί και πέρα την απόφαση την παίρνει η αγορά για να μπορέσει αυτή η διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά. Όπως πολύ σωστά είπατε βέβαια, θα πρέπει να παλύψουμε τα αχρίαστα εμπόδια μεταξύ κρατών μελών, έτσι ώστε να επιτρέψουμε και τις διασυνοριακές ε, συγχωνεύσεις. Και αυτή είναι μια σημαντική διάσταση, αλλά όχι μόνη για να υπάρξει ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο να είναι πιο ποικιλόμορφο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, όντω, ε, οι εποπτικέ αρχέ θέλουν να αποφύγουν την καταστροφή αξίας για τι τράπεζε ε, και τις, ε, και τις απώλειες. Εγώ καλωσορίζω το διαχωρισμό. Θέλουμε να γίνει στο διάλογο να προχωρούμε αναπερίπτωση, ανατράπεζα. Υπάρχουν διάφορε κατηγορίε μη ε, δανείων, τα past due και τα αυτά που ενδέχεται να μην πληρωθούν. Ε, δεν είναι, εφαρμόζουν τους κανόνες πλήρως και όπως πρέπει και οι ίδιες οι τράπεζες και αυτό ορισμένες φορές δημιουργεί περαιτέρω δυσκολίες επιπλέον ε, πρόκειται για μια προσέγγιση αμυγός αναχώρα οι διάφορες κατηγορίες δανείων τώρα ναι βεβαίως ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μεγάλων επιχειρήσεων, διανοπολιτές είναι κάθε περίπτωση διαφορετική εμείς ε, έχουμε εντοπίσει σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες χώρες ε, και όπου υπάρχει έκθεση μη εξυπηρετούν αδάνεια ε, ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να πληρώσουν αλλά δεν πληρώνουν. Δεν πληρώνουν γιατί δεν βλέπουν τον λόγο να πληρώσουν όπως δεν πληρώνουν άλλοι. Είναι στρατηγική δηλαδή ε, εσκεμμένη κάποιον αυτή και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Και ο τελευταίος στόχος θα είναι οι μικροεπενδυτές, λιανοπολιτές, ε, αυτοί που έχουν, ε, παραδείγματος χάρη, ε, απλά μια υποθήκη στο, στην πρώτη κατοικία τους. Εδώ αλλάζουμε τις διατάξεις. Ε, από εκεί που μιλούσαμε για πόλεις που υπάρχουν ήδη, βεβαίως ανακαλύπτονται όταν επιδεινώνονται τα πράγματα, ε, είναι η χειρότερη στιγμή και τώρα όμως μιλάμε πλέον για expected losses, για προσδοκόμενες απώλειες, ε, αναμενόμενες απώλειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι αναμενόμενες απώλειες είναι ε, σωστές, είναι σωστός ο υπολογισμός τους. Εμείς ε, επαναξετάζουμε τα μοντέλα υπολογισμού. Υπάρχουν τράπεζες που ε, υποτιμούν αυτή τη στιγμή ε, τις αναμενόμενες απώλειες. Δηλαδή ενδέχεται οι ελεγκτές για τους λογιστικούς, ε, βάσει κανόνες ε, δεν δίνουν τα σωστά στοιχεία σε εποπτικές αρχές. Αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ευρώπη. Στις περισσότερες χώρες ε, υπάρχει δυνατότητα να πει κάποιος ε, ότι εντάξει αυτό προβλέπει, προβλέπουν λογιστικοί κανόνες, αλλά ε, αν θέλουμε να είμαστε εξασφαλισμένοι μπορούν να προβλεφθούν και περαιτέρω διατάξεις. Μια σειρά από χώρες άλλωστε το κάνουν αυτό στην Ευρώπη. οι χώρε συνήθω οι οποίε τα πήγαν και καλύτερα με την κρίση. Πάντα θα υπάρχει ένα ρόλο. Ε, θα υπάρχει χώρο για τέτοιου είδου περαιτέρω μέτρα. Βεβαίω θα μειωθούν με την εφαρμογή του FRS 9, Έχουμε ακόμα δουλειά μπροστά μας ε, για το αντέντουμ και στις, τα πλαίσια αυτής της ε, ε, αναδιατύπωσής του θα προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη μας και τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου, ε, να δούμε ποια θα είναι η μεταβατική περίοδος για το FRS 9 ε, και τα περαιτέρω προστατευτικά μέτρα. Υπάρχει καταρχήν το τα λογιστικά μέτρα, βεβαίω σίγουρα κανένα, καμιά, ε, καμιά δεν μπορεί να μετρηθεί δύο φορέ. Υπάρχει όμω από εκεί πέρα και τα, και τα περαιτέρω μέτρα, τα προστατευτικά, ε, για συγκεκριμένε ε, συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια και συγκεκριμένες πιστώσεις. Τώρα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, πρόεδρε, τελειώνοντα ε, να πω, ναι, βεβαίω, ε, στείλτε μα τα σχόλιά σα. Εμεί θα τα δούμε, θα τα εξετάσουμε πολύ σοβαρά. Ευχαριστώ πολύ, εκτιμώ ιδιαίτερα την παρέμβασή σα. Ήταν ε, μια ζωντανή, χρήσιμη, θετική συζήτηση. Σας ευχαριστώ και για αυτά που είπατε σχετικά με τα σχόλια που θα λάβετε υπόψη, τα σχόλια του Κοινοβουλίου. Θα γίνει προσπάθεια από ό,τι να βελτιωθεί το κείμενο για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε όλοι. Να έχουμε ένα περαιτέρω εργαλείο για να συνεισφέρουμε σε μια χρήσιμη περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, έτσι ώστε το ε, τραπεζικό μας σύστημα να είναι υγιέστερο και πιο ανθεκτικό. Τώρα για τη θέση σε ισχύ ε, και τη σχετική ημερομηνία, ενδεχομένω είναι ένα σημαντικό στοιχείο και για την αγορά. Πρέπει να το γνωρίζουν και οι εμπλεκόμενοι φορείς. και υπάρχουν και κάποια στοιχεία που χρήζουν βελτίωσης ε, για να εξασφαλίσουμε ε, τον μη αυτόματο χαρακτήρα και την προσέγγιση ένα τράπεζα, όπως είπε η κυρία Νούη. Τα καλωσορίζουμε Αυτό σας ευχαριστούμε πολύ. So, uh, και Κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της Μέσας Διάταξης. Παραμένουμε στον τομέα των ε, τραπεζών, Τραπεζική Ένωση, ετήσια έκθεση για το 2017. Εξετάζουμε το σχέδιο της έκθεσης. σαν Λούνας, ο συγκεκριτής μας. Οπότε έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να ε, κάνω έτσι αν θέλετε τη μετάβαση από τα όσα συζητήσαμε την κυρία Νουή και αυτήν εδώ την έκθεση. Όπως αναφέρατε και εσείς στα συμπεράσματά σας έχουμε τώρα ε, τη νομική γνωμοδότηση σε ό,τι αφορά το παράρτημα για τις ε, ε, κατευθυντήρες γραμμές, πράγμα το οποίο είναι σημαντικό στοιχείο που θα συμπεριλάβουμε και στην έκθεση, σε ό,τι αφορά δηλαδή, την εντολή της Ευρωπαϊκής Σχετικής Τράπεζας και κατά πόσο τελικά αυτά τα στοιχεία ανταποκρίνονται στο βαθμό σημασίας που αποδίδουμε σε αυτό το τομέα. Συμφωνώ μαζί σας Πρόεδρε και για μένα είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα και δεν θέλω να ε, προσθέσω ε, πολλά. Δηλαδή, θα, ενδεχομένως κάποια στιγμή θα πρέπει να ε, συζητήσουμε και την νομιμότητα των δράσεων που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σχέση με άλλα ζητήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έκθεση που εξετάζουμε σήμερα εδώ, δύο λόγια να σας πω. Προσπάθησα εδώ να μην εκφράσω τη δική μου προσωπική άποψη σε αυτό το σχέδιο έκθεση, αλλά προσπάθησα να είναι όσο το δυνατό πιο αμερόληπτη και ουδέτερη γίνεται αυτή η έκθεση. Αυτό ήταν ο στόχο μου. Και γι' αυτό ε, συχνά θα δείτε ότι στην έκθεση αναφέρονται notes, takes notes, δηλαδή σημειώνει η Επιτροπή, έλαβαν υπόψη και ούτω καθεξής. Ε, οπότε ε, γι' αυτό το λόγο ίσως είναι και λίγο ε, γενικόλογη η έκθεση γιατί συχνά αναφέρομαι σε, σε, στοιχεία τα οποία λαμβάνουμε υπόψη μας τα όσα συμβαίνουν. Αλλά και αυτό το έκανα προκειμένου να λάβω υπόψη μου και τα σχόλια που θα κάνουν διάφοροι συνάδελφοι και τα οποία θα εμπλουτίσουν το σχέδιο έκθεσης και δεν νομίζω πως θα υπάρχει έλλειψη σχολείων λαμβάνοντας υπόψη τα όσα συνέβησαν μέσα στο 2017. Τώρα, η έκθεση έχει την ίδια δομή όπως με την περσινή, δηλαδή τρία τμήματα με τα ζητήματα ε, καταθέσεων, ε, την ε, εποπτεία και να πούμε σε ό,τι αφορά την εποπτεία αναφερόμαστε σε ορισμένες από τις περιπτώσεις, υποθέσεις με τις οποίες ασχοληθήκαμε με εξυπηρετούμενα δάνεια, κάποια ζητήματα σύγκλησης σε ό,τι αφορά την οικονομική τεχνολογία, το fintech και εδώ αναγνωρίζουμε τη δουλειά που έχει κάνει το Κόρεβαν Χάουζεν που ανέλαβε τώρα βέβαια καθήκοντα υπουργού στι κατοχώρε. Μετά, στο δεύτερο τμήμα τη έκθεση εξετάζουμε ε, το resolution, την εξηγίαση. Εδώ λοιπόν γίνεται λόγο ε, ε, για την υπόθεση τη Banco Popular και νομίζω πω θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε κάποια στιγμή μια συζήτηση για αυτό το ζήτημα. Ω γενικό σχόλιο να πω ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποφύγουμε μια συζήτηση για την Banco Popular γιατί το πλαίσιό μας τέθηκε σε δοκιμή αν θέλετε με αυτή την περίπτωση, με αυτή την υπόθεση οπότε θα πρέπει λίγο να δούμε ε, τελικά τι, τι λειτουργεί και τι όχι στον τομέα των, ε, των εξηγιάνσεων, δηλαδή προληπτική ανακεφαλαιοποίηση ειδικότερα εδώ μας ενδιαφέρει ε, για μία σειρά από περαιτέρω ζητήματα. Και το τελευταίο τμήμα της έκθεσης περιλαμβάνει ε, τις, ε, τις ασφαλίσεις των καταθέσεων, τα deposit insurances και βέβαια εγώ με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα και το έντις και εδώ με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η σχετική έκθεση ε, της, της ESG γιατί ε, οι συζητήσεις για το ΕΝΤΙ συνεχίζονται ακόμα οπότε ε, εδώ προτείνω σε γενικές γραμμές να κάνουμε αυτό που κάναμε ε, πέρυσι στην περσινή έκθεση δηλαδή οι σχετικές εργασίες να παραπέμπονται εδώ στη δική μας επιτροπή γιατί θα, με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να σε, σεβαστούμε και τα όσα έχει κάνει ο συνάδελφος σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Επίσης Υπάρχει, υπάρχουν και κάποια μικροσφάλματα μέσα στην έκθεση, κάποια αριθμοί δηλαδή που πρέπει να επικαιροποιηθούν, μια ημερομηνία η οποία είναι εσφαλμένη και ούτω καθεξής. Όλα αυτά θα διορθωθούν, αλλά δεν είναι βέβαια ζητήματα ε, που θα μας προβληματίσουν. Προφανώς θα διορθώσουμε και θα τα λάβουμε υπόψη μας και από εκεί και μετά αναμένουμε ενδιαφέροντα σχόλια των συναδέλφων. Ε, σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, η Ντανούτα Χούμνερ ε, που θα πάρει πρώτο λόγο και ότι η για το ΕΛΚ. εκτός μικροφώνου. Δεν ακούγεται κύριε Χρυμπνέ. Oh, direction. So if you want, I move somewhere else. Oh, I can. Okay. Sorry. There is Ελπίζω να λειτουργεί αυτό το μικρόφωνο. Πράγματι λειτουργεί. Ναι. Και ο ε, κύριο Λούνα αποφάσισε να συνεχίσει την ίδια δομή ε, με την περσινή έκθεση έτσι ώστε να έχουμε ε, περισσότερη συνοχή και ανάμεσα στη δική μου έκθεση και αυτήν εδώ και βέβαια προκειμένου να ανταποκριθούμε και στο στόχο ε, που έχουμε θέσει, δηλαδή την βελτίωση του τρόπου με τον οποίο ε, λειτουργεί ο τραπεζικό μα ε, τομέα. Υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που αναφέρονται στην έκθεση, τα οποία είναι γνωστά και τα οποία αναφέρθηκαν και πέρσι προφανώ. Αλλά σε ό,τι αφορά κάποια από αυτά τα ζητήματα, προφανώ θα αποτελέσει έκπληξη το ότι έχουμε διαφορετικέ απόψεις, οπότε αναμένω με ενδιαφέρον τι συζητήσει που θα κάνουμε. Ε, επίσης συμφωνώ ως προς αυτό που αναφέρθηκε ότι δηλαδή πέραν των παραδοσιακών εντό εισαγωγικών ζητημάτων που ε, είχαμε και φέτο. για πρώτη φορά μπορούμε να προβούμε σε μια αξιολόγηση σε ό,τι αφορά ε, την υποθέσει τις πρώτες υποθέσεις ε, και τα διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτές σε ό,τι αφορά δηλαδή την εύρυθμη λειτουργία τη Τραπεζική Ένωση και ποιε είναι οι δυνητικέ βελτιώσει που θα μπορούσαν να γίνουν στην Τραπεζική Ένωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τμήμα τη εποπτεία, ε, θα ήθελα να εστιαστεί η έκθεση λίγο περισσότερο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα εποπτεία των τραπεζών, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του εποπτικού μηχανισμού, του ενίου εποπτικού μηχανισμού του SSM. Και όπω ε, ακούσαμε και σήμερα, ε, θα πρέπει εδώ να εξετάσουμε λίγο και την έκθεση εδώ τη Επιτροπή που δημοσιοποιήθηκε τον Οκτώβριο, γιατί εκεί προέβη πραγματικά σε μια πολύ καλή λεπτομέρεια τρομερή αξιολόγηση των όσων έχουν λάβει χώρα η Επιτροπή και είναι σε γενικέ γραμμέ μια θετική έκθεση. Παρότι βέβαια περιλαμβάνει ταυτόχρονα και μια σειρά από λεπτομερεί συστάσει. Οπότε α εξετάσουμε αυτή την επιτροπή για να δούμε ποιε είναι οι βελτιώσει οι οποίε θα πρέπει να λάβουν χώρα σε σχέση με τον SSM. Επίση, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε το πνεύμα, αν θέλετε, αυτό της ε, ακριβολογίας, αν θέλετε, της έκθεσης, ε, δηλαδή ε, να ασχολούμαστε μόνο με ζητήματα που αφορούν την ε, τραπεζική εποπτεία και τίποτα διαφορετικό. Και άκουσα και τον συνάδελφο Σάντερ ότι δηλαδή ε, πράγματι θέλει να εστιάσει σε αυτά τα ζητήματα και δεν θέλει να προδικάσει ε, ζητήματα που συζητούμε σε ό,τι αφορά την ε, νομοθεσία στο μέλλον, για παράδειγμα το πακέτο για τις τράπεζες, το έντιση και ούτω καθεξής. Οι δικές μου λοιπόν, η δική μου σύσταση είναι ότι ε, σε ό,τι αφορά ζητήματα τα οποία εκκρεμούν ακόμα και συζητούνται ακόμα, ας παραμείνουμε γενικόλογοι σε ό,τι αφορά τις αναφορές που κάνουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις εδώ, δηλαδή τις συγκεκριμένες που αναφέρονται, η δική μου στάση είναι ότι θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ την προστιθέμενη αξία που θα αντλήσουμε ε, από αυτές τις ε, εμπειρίες, από αυτές τις υποθέσεις ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή και το πώς θα βελτιώσουμε την αντιμετώπιση μας στο μέλλον ειδικότερα σε ό,τι αφορά το ζήτημα της, της, ανάμεσα στην εξυγίανση αφενός και την ε, κήρυξη πτώχευσης αφετέρου δηλαδή τις ζημίες σε σχέση με αυτή την πτώχευση την, και να λάβουμε και εδώ υπόψη μας βέβαια την ανακοίνωση σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις αλλά και τα ζητήματα ε, κοινοποίηση, κοινή χρήση των πληροφοριών μεταξύ των ε, φορέων εξηγίαση και των εποπτικών ε, φορέων. Ζητήματα λοιπόν που τα είχαμε συζητήσει και πέρσι και από εκεί και μετά υπάρχει και ένα ζήτημα ε, το οποίο παραμένει και το γεγονό είναι ότι ε, ακόμα βρισκόμαστε στο ίμιση αν θέλετε της διαδικασίας της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα κάποια στοιχεία τα οποία δεν λειτουργούν ακόμα. Οπότε εδώ θα πρέπει ε, η έκθεση να περιλαμβάνει και ε, ε, ένα, να, διαθέτει ένα χαρακτήρα επίγοντος, ότι δηλαδή επίγοντος θα πρέπει να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση. Και εδώ θα πρέπει βέβαια να, ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι θα είναι ισορροπημένη η έκθεση. Δηλαδή ναι με να αναφερόμαστε στον επίγοντα χαρακτήρα των περαιτέρω βελτιώσεων, χωρίς ωστόσο να ξεχνούμε τις θετικές εξελίξεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο του πακέτου που έχουμε συμφωνήσει σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση και τα θεσμικά όργανα αυτής της Ένωσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση αλλά και για την παρέμβασή του. Νομίζω ότι αυτή η επικοδομητική στάση ελπίζω ότι θα ε, συνεχιστεί και στη σύνταξη της έκθεσης. Ε, δύο σχόλια ήθελα να κάνω εισαγωγικά. Καταρχήν καλωσορίζω τη συνέχεια και τη συνέπεια που υπάρχει σε σχέση με τις εκθέσεις του 2015 και του 2016, διότι εδώ έχουμε ε, μια παρακολούθηση και των αξιολογήσεων που έχουμε κάνει στο παρελθόν για να δούμε αν έχει υπάρξει πρόοδος ή όχι ε, για τα διάφορα διακυβευόμενα ζητήματα. Οπότε καλό είναι να ακολουθούμε την ίδια δομή με τα τρία κεφάλαια, είναι κάτι που βοηθάει στην ε, αναγνωσιμότητα του κειμένου. Από πρέπει να δούμε αν υπήρξαν και κάποια γεγονότα σημαντικά που να έλαβαν χώρα το περασμένο έτος και να δούμε εάν αυτά τα γεγονότα αντιμετωπίστηκαν ε, ικανοποιητικά ε, με βάση αυτά που επιθυμεί ο νομοθέτης. Για να έρθω τώρα στην έκθεση αυτή καθ' αυτή. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω την, την έκπληξή μου ε, σε ό,τι αφορά τα εκτιμώντα. Τα εκτιμώντα τα βλέπω τα βρίσκω πολύ αρνητικά. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά εάν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι, θα πρέπει να αναφερθούμε και στην πρόοδο που έχει σημειωθεί. Ακόμα και αν αυτή η πρόοδο δεν είναι επαρκή. Ε, το κεφάλαιο για την εποπτεία τώρα θα είναι χρήσιμο να συμπληρωθεί πιστεύω. Να συμπεριλάβουμε δηλαδή και άλλα στοιχεία εποπτείας όπως ε, η λειτουργία της διακυβέρνησης, ε, των GST, η ανάθεση σε εξωτερικού συνεργάτη, η σχέση μεταξύ των αρχών, η κυβερνοασφάλεια, fintech. Ε, ξέρω βεβαίω ότι δεν γίνονταν να καλυφθούν όλα αυτά τα ζητήματα με βάση το μοντέλο ε, που, έχουν, ε, που ακολουθείται για αυτές τις εκθέσεις. Τώρα, για την εξυγίανση. Ε, πιστεύω ότι θα έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον το κεφάλαιο αυτό. Είχαμε την ίδια την πρώτη περίπτωση εξυγίανσης που βεβαίω θέτει πολλά ερωτηματικά και για την ίδια την εξυγίανση ναι, για το πώς ενεργοποιήθηκε, την αξία της τράπεζας πριν και μετά την εξυγίανση, για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, η επικοινωνία μεταξύ αρχών, αλλά και με τις αρχές άλλων κρατομελών, των οποίων το τραπεζικό σύστημα επηρεάζεται από την εξυγίανση ε, μιας τράπεζας σε μια άλλη χώρα. Να αναρωτηθούμε επίσης για τις επιπτώσεις της εξυγίανσης τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην τραπεζική δομή μιας χώρας, οι ε, επιπτώσεις αυτές είναι θετικές, είναι αρνητικές, είναι επιθυμητές ή όχι. είναι κάπως νωρίς βέβαια, δεν μπορούμε να ε, αντλήσουμε βιαστικά συμπεράσματα από μία και μόνο περίπτωση, αλλά σίγουρα κάτι μπορούμε να μάθουμε ε, για το, από τον Banco Popular και είναι κάτι που θα μας βοηθήσει για το μέλλον. Και τέλος, τελευταίο κεφάλαιο, το EDIS έχω την εντύπωση ότι το μόνο που μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι ότι δεν έχουμε εγγύηση ευρωπαϊκή ε, για τις καταθέσεις και ως τότε όσο υπάρχει αυτό ε, δεν υπάρχει ε, τραπεζική ένωση. Εγώ λέω να ακολουθήσουμε τον κανόνα που συμφωνήσαμε πέρυσι. Να μην προσπαθούν συμβιβασμούς ε, στα γρήγορα για δύσκολα ζητήματα, περίπλοκα, τα οποία εξετάζονται από πολλούς συναδέλφους. Ε, χαίρομαι πάντως για τη συνεργασία που είχαμε. Ελπίζω ότι θα είναι επικοδομητική έτσι ώστε η έκθεσή μας να είναι χρήσιμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τρεμόζα έχει το λόγο από την άλλη Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω εκ μέρους του κυρίου Τιερή Κορνιγέ που δεν είναι εδώ σήμερα. Ο κύριος Κορνιγέ θεωρεί ότι το σχέδιο έκθεσης που έχει υποβληθεί, που υπέγραψε η συνάδελφος Λούνες, είναι ένα καλό σημείο αφετηρίας και θεωρεί ότι αυτή η έκθεση ε, θα μπορούσε να περιλάβει επιπλέον συνεισφορές ο κ. Κορνιγέ θεωρεί ότι ε, στην έκθεση αυτή πρώτα απ' όλα θα πρέπει να υπάρχει μια ρητή αναγνώριση των, του πόσο θετική είναι η Τραπεζική Ένωση. Ε, ε βεβαίως, εντάξει, να το συζητήσουμε το πώς θα το πούμε ακριβώ αυτό, αλλά ε, ο κ. Κορνιγέ θεωρεί ότι πρέπει να είναι σαφές το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από αυτού. Επίσης ε, θεωρεί ότι είναι ένα σημαντικός πυλώνας της νομισματικής ένωσης. Ε, ο κύριος Κορνιγέ είναι υπέρ τρίτου πυλώνα η κοινή ασφάλεια καταθέσεων ε, και πιστεύει ότι σε για να συμβεί αυτό, για να μπορέσει το έντυπο να προχωρήσει, χρειάζεται, χρειάζονται συγκεκριμένε προποθέσει και χρειάζεται εμπιστοσύνη. Έχει κάποιε ανησυχίε ο Κορνιγέ για τι παραγράφου 6, 9 και 10 ε, νομίζω ότι θα έχει χρόνο να τα συζητήσει αυτά στις διαπραγματεύσεις. Και τέλος, ε, έχει την αίσθηση ο κ. Κορνιγέ ότι για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό, ε, ότι αυτό δεν είναι αμυγός εθνικό πρόβλημα. Ε, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος λοιπόν να βρεθεί μια κάποια μορφή σε ευρωπαϊκή λύση. Και ο κ. Κορνιγέ επίσης καλωσορίζει την έμφαση που δίνεται στην έκθεση για την ανάγκη διαφάνειας και καλύτερης επικοινωνίας. Τέλος, έχει γίνει μια αναφορά στην κυβερνοασφάλεια. Πρέπει να, να υπάρξει μια αναφορά στην κυβερνοασφάλεια και στο Brexit στην έκθεση. Αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιέγκας ε, δεν φαίνεται να είναι εδώ, ούτε ο κύριος Ουρτασούν όμως είναι ο κύριος Βάλλη. Παρακαλώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την παρουσίασή του, αν και έχουμε διαφορετικές πολιτικές απόψεις, γιατί η ουσία των προτάσεων δεν τη συμμεριζόμεθα. Δεν συμφωνώ με τις ανησυχίες τις οποίες εξέφρασε σχετικά με τα κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται και με το ενιαίο εποπτικό σύστημα και την συμμετρία είναι σημεία τα οποία υπερβολικά υπογραμμίζονται και επηρεάζουν την πραγματική οικονομία και την πίστοση και δημιουργούν απαιτήσει από τα πιστοτικά ιδρύματα τα οποία δεν επιτρέπουν να βελτιωθεί η ζήτηση, να αυξηθεί η ζήτηση και δημιουργεί και προβλήματα σε σχέση με τα ενεργά δευτέρου και τρίτου επίπεδου. Είναι κάτι που άπτεται και της ρευστότητα των τραπεζικών ε, δομών. Είναι θέματα που θα πρέπει να ληφθούν επιμέρους υπόψη, διότι πολλές φορές γίνεται καταχρηστική χρήση κάποιων στοιχείων της αγοράς και οι τιμές φαίνονται να είναι σε ένα ιδιαίτερα πτυτικό επίπεδο. Στην περίπτωση κρίσης θα ήθελα να σας πω ότι οι τίτλοι ε, σε ρευστό που ε, γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη μη ρυθμιζόμενη αγορά είναι ένας κίνδυνος ε, για τις τράπεζες. Στην ουσία καταστρέφουμε το παραδοσιακό σύστημα δημιουργώντας συνθήκες επιβίωσης των τραπεζικών ίδρυμάτων τα οποία λειτουργούν με αντιλήψεις εντελώς καταχρηστικές και εις βάρος της αγοράς. Πρόκειται για μια αναστροφή ουσιαστικά των πραγμάτων μακράν των συμβιβαστικών τάσεων που θα πρέπει να επιδεικνύουμε τώρα για τις θέσεις του Κοινοβουλίου σε σχέση με την προσθήκη και μετά από την άποψη της νομικής μας υπηρεσίας θα ήθελα στα πρακτικά να εντοπίσουμε κάπως, να σημειώσουμε ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας από τη μία και οι διακανονιστικές και νομοθετικές ικανότητες του Κοινοβουλίου από την άλλη. Για τα bail-in είμαστε κατά σαν σύστημα, γιατί πιστεύουμε ότι δεν είναι ουσιαστικό βήμα προόδου για την Τραπεζική Ένωση ε, υπάρχει η έννοια της λεγόμενης Universal Bank καθολικής, καθολικού ενδιαφέροντος ε, τράπεζας και δημιουργείται σύγχυση με επενδυτικές τράπεζες κτλ. Θα πρέπει λοιπόν και οι καταθέτες στα πλαίσια της Τραπεζικής Ένωσης και οι φορολογούμενοι να ε, είναι σε θέση να διασώσουν τις τράπεζες, οι οποίες τράπεζες όμως υφίστανται πάρα πολλές πιέσεις σε επίπεδο χρηματοπιστωτικών αγορών και σε καμία περίπτωση δεν είναι ρόλος του φορολογούμενου να δίδει εγγυήσει για παράλογες εμπορικές πρακτικές στον τομέα των πρακτικών. Τώρα, βλέπω ότι οι εγγυήσει που δίδονται στα διάφορα κράτη-μέλη είναι διαφορετικού επίπεδου. Ε, τα διάφορα κράτη έχουν χρησιμοποιήσει δύσεις για να βοηθήσουν τα τραπεζικά του στοιχήματα τα τελευταία χρόνια και να καλύψουν κάποιες ε, θα έλεγα καταστάσεις οι οποίες δεν είναι ξεκάθαρες γιατί από το 11 μέχρι το 13 χρησιμοποιήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια στο γερμανικό σύστημα, στο ολλανδικό σύστημα και άλλες χώρες στην Ιταλία σαν παράδειγμα το έκαναν αργότερα και οι δυσκολίες είναι τεράστιες και γι' αυτό απαιτείται να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε αυτήν την συμμετρία που είπα. Τώρα για τον τρίτο πυλώνα υπάρχει ανάγκη να δώσουμε μένα από τη μία προστασία στους ε, καταθέτες, στους αποταμιευτές να υπάρξει δυνατότητα ε, διαμήρασης του κινδύνου μέσω του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων και ταυτόχρονα στο εσωτερικό ε, των διαφόρων συνταγματικών αρχών, ε, μάλλον χαρτών στις διάφορες χώρες υπάρχει το δικαίωμα στην αποταμίευση και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει και η δυνατότητα σε περίπτωση ε, κρίσης ε, να προστατεύεται η αποταμίευση και να μην δημιουργούνται προβλήματα στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος. Ελπίζω να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σωστά με τον εισηγητή και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιες ε, θέσεις κοινέ, αν και εξακολουθούν να αφίστανται οι θέσεις μας τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω την αίσθηση ότι θα ήταν καλό να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο καταρχάς να είναι λειτουργικό. Ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέψει στην πολιτική μας ομάδα να παίξει ε, και τον ρόλο της ως εισηγητρίας στην συγκεκριμένη περίπτωση, ανεξάρτητα από αυτά τα οποία προτείνει η κυρία Μπέρες. Τώρα ο μηχανισμός αυτός που είναι το αντικείμενο της έκθεσης, καλό θα είναι να επανέλθουμε λίγο στην έκθεση του Λούνς. Εγώ έχω μια πολύ προσωπική ίσως άποψη πάνω σε αυτό και δυστυχώς αυτά τα οποία λέγει είναι πολύ γενικόλογα και δεν μας δίνουν πάρα πολλές δυνατότητες παρέμβασης. Γίνονται πολλές αναφορές στα θετικά στοιχεία, αλλά δεν γίνονται επαρκείς αναφορές στα προβληματικά στοιχεία και ιδιαίτερα σε σχέση με τις κατεξουσιοδότηση πράξη. να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε περισσότερο σε σχέση με το SSM. Λοιπόν, λαμβάνουμε υπόψη την στάση της Κεντρικής Τράπεζας, λαμβάνουμε υπόψη τον ρόλο που έπαιξε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα σε σχέση με την Banco Popular. Θα έπρεπε να το συζητήσουμε ακόμα περισσότερο αυτό, αναφέρθηκε και η κυρία Νούη σε αυτό. Δόθηκαν κάποια παραδείγματα και για άλλες τράπεζες, όπως σαν παράδειγμα την Banca Veneto στην Ιταλία, Οπότε καλό θα είναι να προσπαθήσουμε να περάσουμε σε ένα υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε άλλου τύπου συμπεράσματα σε σχέση με τις προτάσεις οι οποίες γίνονται. Είναι λίγο παράδοξο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η τράπεζα η Ιταλική Monte dei Paschi di Siena όπου υπήρξε λήψη μέτρων για την προστασία των καταθετών της τράπεζας αυτής σε προληπτικό επίπεδο. Είναι μια έκθεση που παρουσιάστηκε στις 20 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος κύριε Λούνες. Από τότε έχουν υπάρξει όμως εξελίξεις σε χρηματιστηριακό επίπεδο για την Monte Dei Paschi και πολλοί καταθέτες και επενδυτές έχασαν χρήματα. Οπότε διαρωτώ με τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Οι επενδυτές λοιπόν σήμερα δεν έχουν εμπιστοσύνη σε σχέση με τον μηχανισμό ο οποίος λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και κυρίως στην Ιταλία. Σχετικά τώρα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η πρόταση η οποία έγινε δεκτή από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου χαιρετίστηκε από την ε, πλειοψηφία των συναδέλφων Κάποιοι από τους συναδέλφους όμως και ο κύριος Λούνες καταψήφισε την πρόταση όπως και άλλα μέλη του της ομάδας των συντηρητικών. Παρ' όλα αυτά ο εισηγητής καταφέρνει και κάνει κάποιες προτάσεις οι οποίες είναι θα έλεγα λίγο διαφοροποιημένες και βλέπω εδώ ουσιαστικά ότι οι τράπεζες αλλά και τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αν δεν το κάνουν αυτό δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για άλλα θέματα όπως οι λεγόμενες δευτερεύουσες ε, υποχρεώσεις και ευθύνες. Τέλος, δύο επιπλέον στοιχεία για τα ε, ε, ευρωομόλογα. Λέει η έκθεση takes note, λαμβάνει υπόψη σημειώνει. Αυτό δεν λέει τίποτα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε τις απόψεις σας. Εγώ είμαι ιδιαίτερα σκεπτικιστής και θα, γι' αυτό και θα περίμενα από πλευράς του εισηγητή ακόμα περισσότερο σκεπτικισμό επίσης. Νομίζω ότι είναι ένα γλίστριμα προς μια κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα οδηγήσει στην Δημοσιονομική Ένωση κάποια στιγμή και γι' αυτό θα έπρεπε να ασκηθεί σκληρή κριτική. Το ίδιο ισχύει και για το έντις και εδώ είμαι ιδιαίτερα σκεπτιστική σε σχέση με το έντις. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που θα εξυπηρετήσει το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο σαφείς και πιο ξεκάθαροι. Περιμένουμε βέβαια την έκθεση έντις, αλλά η διατύπωση και η περιγραφή των κινδύνων που δημιουργεί το σύστημα αυτό θα έπρεπε να περιγράφεται με σωστότερο τρόπο προσωπικά θα ήθελα να πάρω μέρος στην σύνταξη μιας έκθεσης για την ε, Τραπεζική Ένωση η οποία είναι αναμενόμενη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σκοβούρ. Ah. Thank you, Senor Presidente. Um, Madam Ευχαριστώ. Πρόεδρε, η κυρία Νόη μα είπε σήμερα ότι η οικονομία βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Εγώ δεν είμαι πεπισμένο ε, και ε, μετά από κάποια χρόνια που έχω εμπειρία στον ε, τομέα της των χρηματοπιστωτικών αγορών βλέπω ότι όταν κάτι πάει καλά επίκειται κάτι άσχημο. Οπότε σε ό,τι αφορά τη σχετική πολιτική σε αυτό το τομέα, εδώ έχουμε ένα θεμελιώδες, και, ε, ένα θεμελιώδες πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διαονίζεται πάντοτε και είναι ο λόγος για τον οποίο ε, αποχωρεί και το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι δηλαδή ότι υπάρχει πάντα ενιαία λύση πάντοτε για όλους και υπάρχουν ε, και βέβαια καταστροφικές αλυσιδωτές αντιδράσεις. Δηλαδή εάν ένας ε, αποτυχάνει σε κάτι όλοι αποτυχάνουν. Από εκεί και μετά δεν υπάρχουν και αξιολογήσεις αντικτύπου σε ό,τι αφορά αυτή την ένωση. Οπότε ε, δημιουργείται ένα συστηματικό κίνδυνο για τις τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και γενικότερα για την οικονομία. Αυτές είναι οι ανησυχίες λοιπόν που θα ήθελα να τονίσω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που να, ζητήσουν, να ζητούν το λόγο. Οπότε ο συνάδελφο Έλβας, ε, ναι, σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας και θα λάβω υπόψη μου όλες αυτές τις τροπολογίες και εγώ προφανώς θα, θα ε, υποβάλλω τροπολογίες ώστε να ε, αντικατοπτρίζονται ε, τα όσα συζητούνται εδώ η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, να απευθυνθώ πολύ σύντομα στον κύριο Ασεμάς και να πω ότι Προφανώς μπορώ να συμπεριλάβω τροποποιήσεις μέσα σε αυτό το ε, σχέδιο έκθεσης, αλλά σε ό,τι αφορά τις δικές σας τροπολογίες, μετά από τις συζητήσεις που κάναμε με το ENF, ε, εντάξει, αναλάβετε δράση εδώ. Ε, γιατί βλέπουμε ότι σε ορισμένους πατέλους μπορούμε να επιτύχουμε κάτι πάρα, πάνω, σε, σε άλλους τομείς δεν ε, υπάρχει τόσο μεγάλη συμφωνία, αλλά ε, εντάξει, βλέπουμε ότι έχει επανειλημμένα αξιοποιηθεί αυτή η πολιτική της ε, άδεια κάρεκλας. Ε, πάντως, υποβάλλετε τις τροπολογίες σας. Ε, καλώς λέω πρόεδρος, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Έως 21 Νοεμβρίου υποβολή τροπολογιών, εξέταση των τροπολογιών 7 Δεκεμβρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 24 ή 25 Ιανουαρίου, με στόχο την ψήφιση ε, του σχεδίου της έκθεσης στην Ολομέλεια στις 2 ε, Φεβρουαρίου. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ τον εισηγητή και τους σχέδες και όσο συμμετείχαν στη συζήτηση και περνάμε τώρα στην ετήσια έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού. Ε, εισηγητής εδώ ο κύριος Τρεμόζα, έχετε το λόγο. Dear colleagues. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί πρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για δεύτερη φορά είμαι συγκητής αυτής της έκθεσης για την πολιτική ανταγωνισμού και κατά τα τελευταία 8 χρόνια είμαι ούτε συγκητής τη πολιτική μου ομάδας, επανειλημμένα σχέση με αυτό το ζήτημα. Οπότε πραγματικά μου αρέσει η σύνταξη αυτών των εκθέσεων γιατί ε, μας δίνουν ε, μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Επιτροπή μας. γνωρίζω καλά ότι πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας, κατά συνέπεια όχι νομοθετικού χαρακτήρα. Άρα ο, το καλύτερο μήνυμα το οποίο μπορούμε να διαβάσουμε στους πολίτες μας και στην Επιτροπή είναι ένα μήνυμα το οποίο θα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη δυνατή ε, πλειοψηφία ε, στην Ολομέλεια κατά την ψήφιση ε, αυτής της έκθεσης. Οπότε ο στόχος μου και πάλι θα είναι αυτός, να έχουμε το μεγαλύτερο ε, τη μεγαλύτερη ε, δημοκρατική ομοφωνία και δημοκρατική εντολή στο πλαίσιο αυτή τη έκδοση. Και γι' αυτό ακριβώ θα λάβω υπόψη μου όλε τι ε, πτυχέ και όλε τι απόψει, προκειμένου να κάνουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα σχόλια στην Επιτροπή, στα οποία θα μπορέσει εκείνη να δώσει συνέχεια κατά τα επόμενα χρόνια. Κατά την πρώτη λοιπόν αυτήν ανταλλαγή απόψεων που θα κάνουμε θα σας αναφέρω κάποια στοιχεία τα οποία έχω συμπεριλάβει στην έκθεσή μου και τα οποία βέβαια μπορείτε να τροποποιήσετε με σας. Όπως κάναμε λοιπόν κατά τα τελευταία έτη, ε, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, παράσχει τα απαραίτητα κονδύλια στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Γιατί όπως ε, γνωρίζετε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού είναι αρμόδια για μία σειρά για υποθέσεις έναντι πολυεθνικών γιγάντων και αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μόνο δικηγόρους ε, και άλλους αλλά ε, και μηχανικούς στον τομέα της, της προηγμένης τεχνολογίας ούτως ώστε να μπορεί να, να, να εξετάζει το τι συμβαίνει σε αυτούς τους τομείς. Άρα λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίζει να υποστηρίζει όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια ε, ένα τέτοιο αίτημα για περισσότερη χρηματοδότηση Γενικής Διευθύνσης Ανταγωνισμού. Επίσης στην έκθεσή μου ζητώ από την Επιτροπή να επαληθεύσει ότι εθνικές αρχές ανταγωνισμού, NCS δηλαδή, διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς ε, και ε, πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό τους ώστε να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους στα διάφορα κράτη-μέλη. Είναι δηλαδή μια ανάγκη που αυτή θα πρέπει να καλύπτεται και νομίζω πως ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε από αυτού. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα όσα επιτυχάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν το ίδιο αντίκτυπο και δεν Επιτυχάνουμε με τον ίδιο τρόπο στα κράτη-μέλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, τα ζητήματα αδικία, σε ό,τι αφορά φορολογικά ζητήματα, ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα ε, και με απασχολεί ειδικότερα σε ό,τι αφορά το φορολογικό ανταγωνισμό, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι η βασική αρχή είναι όλοι οι συμμετέχοντες στην οικονομική δραστηριότητα θα πρέπει να καταβάλουν με δίκαιο τρόπο το δικό τους μέρος μας εφόρους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι ε, συμβαίνει συγκεκριμένα σε ορισμένε περιπτώσει, όπω για παράδειγμα τη Amazon στο Λουξεμβούργο. Οπότε θέλω να ξεκινήσει μια συζήτηση σε σχέση με αυτό το ζήτημα, γνωρίζοντα ε, πολύ καλά πω οι φορολογικέ πολιτικέ παραμένουν εθνική αρμοδιότητα σε πολιτικέ. Α μιλήσουμε όμω για αυτό το ζήτημα, γιατί πολλοί πολίτε ζήτησαν την άποψη του Κοινοβουλίου σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τώρα την Google. Υπάρχει εδώ ένα γεγονός. Υπάρχει δηλαδή μία απόφαση της ε, ε, Επιτροπής, ε, θεωρείται δηλαδή αυτό το comparison service της Google παράνομο και κατά συνέπεια τώρα έχουν επιβληθεί συγκεκριμένε υποχρεώσεις. Αυτό είναι λοιπόν το γεγονό, αυτό που έχει λάβει η χώρα. Οπότε, καλό την Επιτροπή να παρέμβει και σε άλλους τομείς ε, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τις αναζητήσεις για ταξίδια αλλά και τις τοπικές αναζητήσεις όπου η Google ε, κάνει κατάχρηση ακριβώς της ηγετικής ε, θέσης στην αγορά. Οπότε καλούμε να γίνει αυτή η εξέταση όπως και η εξέταση του λογισμικού Android. Επίσης απευθύνουμε μία πρόσκληση απέναντι σε όλους τους ευρωβουλευτές να καλέσουμε την, και τον Γενικό Διευθυντή της ΕΣΥΟ και να συμμετάσχουν για παράδειγμα σε, ε, στις ακροάσεις ε, των ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών ΕΚΟΝ αλλά και τη ΙΜΚΟ γιατί ε, μια τέτοια ακρόαση θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και θα μπορούσε να την παρακολουθήσουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε. Αυτή λοιπόν η συζήτηση ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να βρεθούν εδώ μαζί μα στο Κοινοβούλιο στι Βρυξέλλε και να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα πρόστιρα, μιλάμε για σημαντικές επιπτώσει. οπότε ε, θα μπορούσαμε να περάσουμε με αυτόν τον τρόπο ένα εμφατικό μήνυμα. Εάν δηλαδή συγκεντρώναμε ε, την συνένεση πολλών συναδέλφων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς μια τέτοια ακρόαση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τομέα της αεροπορίας, εδώ ε, ζητούμε από την Επιτροπή να εφαρμόζει αυστηρά και ομοιόμορφα τους ε, σχετικούς κανόνες σε όλες τις αεροπορικέ επιχειρήσει, γιατί έχουν προκύψει κάποια ε, προβλήματα με την Αλιτάλια και την Air οπότε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή και αυτή η δυνατότητα. Επίση, ε, χαιρετίζουμε την αναθεώρηση του κανονισμού 868 του 2004 σε ό,τι αφορά την, ε, τον, το θεμητό ανταγωνισμό και την εξάλληψη των καταχρηστικών πρακτικών. Ε, θεωρώ ότι ε, είναι σημαντικό αυτός αυτή η πτυχή της διαφάνειας στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού είναι απαραίτητο ώστε να υπάρχουν ίσοι όροι του παιχνιδιού. Σε ό,τι αφορά τώρα τα, τους αερολιμένες και την αποτελεσματικότητα των κρατικών ενισχύσεων θεωρώ πω όταν χρησιμοποιούνται δημόσια κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την επένδυση σε υποδομέ, ε, θα πρέπει να λαμβάνει η χώρα μια ανάλυση κόστους αποτελέσματος η οποία θα πρέπει να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να επιτρέπεται η χρηματοδότηση αυτή. Και επίσης καλούμε την Επιτροπή να συντάξει ένα ε, κατάλογο αυτών των, ε, των κόστων, cost airports γιατί ε, γιατί γνωρίζετε πως έχει γίνει λόγο σε διάφορα θεσμικά οργανά για αυτά τα ενεργολουμένων, οπότε ε, θεωρούμε πως ε, καλό θα ήταν η Επιτροπή που έχει τις σχετικές πληροφορίες να συντάξει ένα σχετικό κατάλογο. Τέλος, σε ό,τι αφορά το τομέα της, της γεωργίας και ειδικότερα των αγροτικών τροφίμων, θεωρώ πως θα ήταν ενδιαφέρον να αναλύσουμε εδώ και να ζητήσουμε από την Επιτροπή να διερευνήσει το πώ η έλλειψη ανταγωνισμού, η απουσία ανταγωνισμού σε ορισμένα τμήματα τη Αλυσίδα τροφίμων θα μπορούσε να έχει επιπτώσει ή έχει επιπτώσει στι ε, τιμέ των αγροτικών τροφίμων και πώ επηρεάζει και το εισόδημα των ε, παραγωγών αγροτικών τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λοιπόν είναι τα κυριότερα στοιχεία που έχω συμπεριλάβει στην εκθεσή μου και αναμένω τα σχόλια των συναδέλφων και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο για το ΕΛΚ, ο κύριο Στολίχη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τι να πω, εάν δείτε το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα του ανταγωνισμού, χωρίς δισταγμό μπορεί να πει κανείς ότι είναι εξαιρετική η δουλειά αυτή. Ίσως η φετινή έκθεση η ετήσια για τον ανταγωνισμό να πρέπει να είναι πιο σύντομη σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ο εισηγητής έχει κάνει καλή δουλειά. Εκτιμώ ε, την υποστήριξη της ανεξαρτησίας της Κομισιόν αλλά και των εθνικών αρχών στον τομέα του ανταγωνισμού αυτό μπορεί να γίνει όπως λέει πολύ σωστά ο εισηγητής, εξασφαλίζοντας ότι θα υπάρχουν οι απαραίτητοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι ε, που χρειάζονται αυτές οι αρχές. Εκτιμώ επίσης ε, την τακτική επαφή με τους ε, επιτρόπους επιφορτισμένους με τον ανταγωνισμό, εδώ στην Επιτροπή Εκών εννοώ, αλλά και στο Κοινοβούλιο γενικότερα. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τη σε βάθος ανάλυση ε, στη, για τις ε, πρακτικές που αντιβαίνουν τον ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά τα φορολογικά πλεονεκτήματα που μπορεί να λύσει κάποιος, οι κανόνες περικρατικών ενισχύσεων πρέπει να εφαρμόζονται ε, και για τις ε, φοροαπαλλαγές και για οποιαδήποτε άλλη μορφή ε, ενίσχυσης. Και βεβαίως να υπάρχει και ανάκτηση της κρατικής ενίσχυσης όταν αυτή είναι ασύμβατη. Να επιστρέφεται δηλαδή. Θα ήθελα βεβαίως να έχω την αντίδραση του εκπρόσωπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γύρω από κάποια ζητήματα. Το πρώτο αφορά κάτι που αναφέρεται και στην έκθεση. Στην έκθεση υποβάλλεται μια πρόταση να θέσουμε κάποιους στόχους ε, χρονικούς σε ό,τι αφορά τις έρευνες ε, για, τις, ε, για των τραστ όπως και για τα επίσημα μέτρα που παίρνονται δηλαδή θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το αίτημα που έχει προσθέσει ο εισηγητής στην έκθεση. Επίσης στην έκθεση υπάρχει μια πρόταση έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μελέτες για τη συγκέντρωση των τραπεζών ε, που έλαβε χώρα μετά από την οικονομική κρίση. Ίσως να είναι καλή ιδέα να πω ότι η κατάσταση βεβαίως διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στη χώρα μου, παραδείγματο χάρη, στη Ρουμανία έχουμε πολλές τράπεζες, υπερβολικά πολλές τράπεζες και η διαδικασία συγχώνευσης ε, ε, αγορά, ε, εξαγοράς είναι εν εξελίξη. Σε κάποια άλλα κρατημέλη σε κάποια κρατημέλη μάλλον είναι θετικό, θετική συγκέντρωση και οι συγχωνεύσεις. Αυτή η διαδικασία άλλωστε ε, εποπτεύεται από τις αρχές ανταγωνισμού των χωρών αυτών. Θα ήθελα να ξέρω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για αυτή την πρόταση και κάποια άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαφάνεια. υπάρχει εδώ μια δέσμευση ότι για κάθε ενίσχυση που ξεπερνάει το μισό εκατομμύριο ευρώ, τις 500.000, υπάρχει υποχρέωση στα κράτη-μέλη αυτό να δημοσιεύεται, να δημοσιοποιείται, να είναι διαφανής διαδικασία. Μήπως είναι ψηλό όμως αυτό το όριο, 500.000. Για μια πλούσια χώρα, εντάξει μπορεί να μην είναι μεγάλο το όριο, αλλά για άλλες δεν είναι λίγα λεπτά. Ίσως θα πρέπει να προβλέπετε ένα χαμηλότερο όριο. Τελευταίο που θα ήθελα να θέσω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπλόκαρε τη συγχώνευση μεταξύ της Deutsche Bank και του London Stock Exchange. Αυτή η απόφαση πάρθηκε πριν το Brexit. Το Brexit επηρεάζει αυτή την απόφαση. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το Brexit θεωρεί ότι να μπλοκάρουμε αυτού του είδους συγχωνεύσεις είναι η σωστή απόφαση. Ξεκολουθεί να είναι η σωστή απόφαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Άλφρετ Σαν τώρα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Να συγχαρώ τον κύριο Τρεμόσα Υπάρχουν σημεία προσυζήτηση που θα βελτιώσουν την έκθεση αυτή. Αν και κάποιοι θα μπορούσαν να το κατηγορήσουν ότι εκφράζει πολύ φιλελεύθερες απόψεις στην πρότασή του. Είναι σαφές ότι το ένα μέγεθος για όλες τις περιπτώσεις είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Οι κρατικές παρεμβάσεις σε ορισμένα σενάρια είναι καλοδεχούμενες. Και στο πλαίσιο αυτό καλύπτονται οι επιδοτήσεις ή κρατικές σε τομείς όπως οι μεταφορές και η ενέργεια. Είναι σαφές λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει και την παροχή ενέργειας, την εύρυθμη λειτουργία και τις μεταφορές. Οι κρατικές επιδοτήσεις βέβαια προς τις αεροπορικές επιχειρήσεις είναι κάτι το οποίο δεν είναι απόλυτα εξισορροπημένο σαν πρακτική. Η αναδιάρθρωση πολλές φορές των επιχειρήσεων αυτών απαιτείται η κατάργηση αριθμού πτήσεων προς ε, ε, απότερες περιφέρειες όπως επίσης και περιοχές με πολύ χαμηλή ε, κίνηση. Θα πρέπει επίσης να ελεγχθούν οι εργασιακές σχέσεις που παρέχουν στο προσωπικό τους, που επιβάλλουν μάλλον στο προσωπικό τους οι, ε, ε επιχειρήσεις, αεροπορικές χαμηλού κόστους. Τώρα για το άνοιγμα των, ε, των, για την ιδιωτικοποίηση των λιμένων, αερολιμένων κτλ. πολλές φορές ε, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα κρίσιμο, αλλά μερικές φορές ε, για τις απότερες ε, περιφέρειες όπως επίσης και τις νησιωτικές περιοχές είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αφήσουμε πλήρως στην λειτουργία της αγοράς από μόνη της. για τις εθνικές αρχές εποπτείας είναι σωστές οι προτάσεις του εισηγητή αλλά να υπογραμμίσουμε και την σημασία της αρχής της επικουρικότητας. Τώρα το Google είναι στην επικαιρότητα. Είναι όμως κάτι το σαφές στον ψηφιακό κόσμο ότι ισχύει σήμερα γιατί αλλιώς τότε είναι σαν να αγνοούμε τον ελέφαντα που είναι ήδη μέσα στο δωμάτιο. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα και να επιτρέψουμε στην καινοτομία να ανθίσει. Είναι κάτι το οποίο βέβαια δημιουργεί αβεβαιότητα ε, προς όλες τις κατευθύνσεις ε, και ένα θέμα το οποίο επανέρχεται πάρα πολύ συχνά είναι η σωστή κατανομή ανθρώπινων πόρων και χρηματικών πόρων ε, σε τομείς όπως η εποχιακή εργασία κτλ. Και αυτό ισχύει και για τον τομέα της ψηφιακής οικονομίας, όπου απαιτούνται εργαζόμενοι με υψηλή εξειδίκευση. Είναι κάτι το οποίο βέβαια θα πρέπει να δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ανάγκες που έχει σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων, δεν μπορεί να είναι κριτής και κρινόμενος ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ. Τέλος, το αίτημα της ε, πρότασης ε, για την έλλειψη ανταγωνισμού σε τμήματα της, τροφιμικής, της διατροφικής συγγνώμη, αλυσίδας είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στους παραγωγούς και θα πρέπει να επανεξεταστούν και τα επιμέρους προβλήματα των ε, αγροτών μικρής κλίμακας. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Λούνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον φίλο Τρεμόσα. Θέλουμε να συνεχίσουμε τον διάλογο. Ξέρουμε ότι οι Καταλωνοί είναι υπέρ του διαλόγου, είναι υπέρ της ελευθερίας έκφρασης και σε περιπτώσεις ανταγωνισμού ανάμεσα σε επιχειρήσεις, περιφέρειες, κράτη-μέλη και γι' αυτό θα συνεχίσουμε νομίζω με επιτυχία τον διάλογο οραμών. Τώρα για το συγκεκριμένο θέμα θα ήθελα να περιοριστώ σε ορισμένες παρατηρήσεις. Φορολογία καταρχάς. Η φορολογία είναι ε, κατεξοχήν αρμοδιότητα των κρατών μελών και ελπίζω στο μέλλον και περιφερειών και γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω στον εισηγητή να συγκεντρώσει την προσοχή του στον ανταγωνισμό και να μην μπει ε, σε θέματα φορολογίας. Θα συμφωνήσω βέβαια ότι κάποιες ε, επιδοτήσεις ε, κρατικές οι οποίες είναι εναντίον της έννοιας του ανταγωνισμού στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά. Δεύτερον, το Κοινοβούλιο οφείλει να έχει λόγο στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής για τον ανταγωνισμό, αλλά προτείνω να μην κρίνουμε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και περιπτώσεις. Γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Uh, και θα πρέπει να σταματήσουμε να ονοματίζουμε τις μεμονωμένες επιχειρήσεις και δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να χτυπάμε την Google συνεχώς. Έτσι κι αλλιώς θα γίνει κάποια συζήτηση όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Τώρα για τον σημαντικό ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στα πλαίσια της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς είναι θέμα το οποίο παραδοσιακά μας απασχολεί Ζητάμε λοιπόν να ανακατανείμει τους πόρους τους οποίους έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε η υπηρεσία αυτή της Κομισιόν να έχει περισσότερους ανθρώπους να κάνουν τις έρευνες που απαιτούνται και να μην δαπανώνται οι πόροι αυτοί σε άλλες γενικές διευθύνσεις που έχουν μικρότερη σημασία. Τέταρτον, θα μπορούσαμε στα πλαίσια της έκθεσης αυτής να λάβουμε υπόψη μας ε, και τα προγράμματα προμηθειών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ε, Διοίκησης και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να δούμε πώς ε, κάνουν τις επιλογές τους όταν προχωρούν στην αγορά ομολόγων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει στο μέλλον. Θέλω λοιπόν να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ακριβώς στα πλαίσια του ελεύθερου καταλανικού πνεύματος για τον διάλογο και την ανεξαρτησία. Σας ευχαριστώ πολύ. Η λόπετε Μέχο. Ευχαριστώ να ευχαριστώ καταρχήν τον εισηγητή για το έργο του. Ε, συμφωνώ με τις βασικές προτεραιότητες όπως η καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής, ε, ε, η εξερεύνηση των μεγάλων ψηφιακών μονοπωλίων όπως η Google ή η Amazon. Ε, η Κομισιόν προχωράει βεβαίως προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι αργή η πρόοδος, είναι αργές οι έρευνες και προχωρούν μόνο με βάση την πολιτική πίεση και την πίεση των μέσων ενημέρωσης. Θέλουμε πιο μεγάλη ταχύτητα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημαντικά ζητήματα όμως σε ό,τι αφορά την πολιτική ανταγωνισμού. Ε, πρώτα απ' όλα η γεωργία. Ε, έχουν υποθεί κάποια πράγματα, αλλά εδώ υπάρχει μια ενοποίηση των παραγωγών, ε, τους πόρους, ε, τα λιπάσματα, ε, συγχώνευση της Μοντσάντο με της Bayer, η, η Down Depont με μια κινέζικη εταιρεία. Δεν μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε η γεωργία να πέσει στα χέρια των μεγάλων πολυεθνικών και να μην έχουν πρόσβαση στη γνώση οι γεωργοί. Εδώ χρειάζεται αντίδραση της Κομισιόν. Στο άλλο άκρο τώρα, στην άλλη της, ε, της γεωργικής αλυσίδας, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σειρά από εργαλεία ελέγχου της τιμής των σιτηρών, του κρέατος, του γάλακτος κτλ. Ε, και νομίζω ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία τώρα ε, για να, υπάρξει, να, να λάβει δράση κατά των ενδιάμεσων, κατά των μεσαζόντων, αυτά των κερδοσκόπων που κερδοσκοπούμε τις τιμές εις βάρος όλων των υπολείπων. Θα πρέπει επίση η Κομισιόν να επαναξετάσει κάποιε από τι αποφάσει που έχει πάρει στον ενεργειακό τομέα, έτσι ώστε να είμαστε πιο συνεπεί και να συμπληρώσουμε τη μετάβαση προ ε, μια βιώσιμη, κυρίαρχη και δημοκρατική ε, προσέγγιση. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ε, τους μηχανισμούς ε, της ε, υπερ, υπερβολικής δυνατότητας ε, βλέπουμε ότι αυτό είναι υπέρ τη πετρελαϊκή βιομηχανία ε, και κατά των νέων πηγών ενέργειας. Ε, ενώ υπάρχει το υπερβολικό κόστος για το moratorium, παραδείγματο χάρη για τα πυρηνικά, οι υδροκριτικέ εταιρείε. Τέλος, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να φροντίζει να υπάρχει μια, σωστή λειτουργία της αγοράς, αλλά όχι να αποσαρμολογήσουμε μια σειρά από οργανισμούς που λειτουργούν σωστά μετά την, ε, ε την αποβιομηχανοποίηση, ε, τα προβλήματα στον τομέα των ε, μεταφορών, των σιδηροδρομικών. Ο ρόλος της Κομισιόν είναι αμφίσιμος και συχνά οδηγεί σε κοινωνικό ντάμπινγκ χωρίς πραγματικά ωφέλη για τους καταναλωτές και τους χρήστες ενώ ε, τα ολιγοπόλια που δημιουργούνται προχωρούν ενόχλητα. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω πρόσωπο από τους πράσινους. Ωραία. Από την ΙΕΝΕΦ ούτε την EFDD. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Όχι. Ο εισηγητής έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά μόνο να ευχαριστήσω για την εισφορά. Ε, κύριε Στολογιάν, καλό θα ήταν να συζητήσουμε βεβαίω όλοι εμεί για το μέλλον του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη. Διότι ανησυχώ για τι αποκλήσει που διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια. Από ό,τι φαίνεται σε κάποια κράτη-μέλη στον Νότο υπάρχει μια σαφής προτίμηση μόνο, να υπάρχουν μόνο τρεις μεγάλοι παίχτες, τρεις μεγάλες τράπεζες ε, στην Ισπανία οι τρεις μεγάλες τράπεζες αυτές ε, καλύπτουν 70% όλης της τραπεζικής πίστης. Αυτό ε, δείχνει ότι αυτές οι τράπεζες ε, είναι εξαιρετικά συστημικές. Εάν μία από αυτές τις τράπεζες αντιμετωπίσει πρόβλημα, θα υπάρξει πρόβλημα με την πίστη ολόκληρη της, χώρα, ολόκληρη της χώρας. Εγώ νιώθω πιο ασφαλής σε ένα μοντέλο όπως το γερμανικό, όπου υπάρχει μια ομάδα μεγάλων τραπεζών, αλλά υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο και πυκνό δίκτυο εκατοντάδων μικρών και μεσαίων τράπεζων αποταμίευσης. Η Deutsche Bank, παραδείγματος χάρη, που αντιμετώπισε προβλήματα τα τελευταία έτη, εκπροσωπεί μόνο το 6% της συνολική πίστη στη Γερμανία. Εάν προκύψει πρόβλημα με την Deutsche Bank, δηλαδή οι γερμανικές αρχές μπορούν να το διαχειριστούν. Γι' αυτό λοιπόν ανησυχώ ε, για αυτό που συμβαίνει με αυτή τη συγκέντρωση σε κάποια κράτη-μέλη. Ε, είναι διαφορετική η προσέγγιση από ό,τι φαίνεται σε κάποιες βόρειες χώρες και τα αποτελέσματα θα είναι επίσης διαφορετικά όταν θα προκύψει μια νέα οικονομική κρίση ή αν έχουμε κάποιο εξωτερικό σοκ. Πάντω ευχαρίστω να συμπληρώσω με τον κύριο Στρό γιατί ξέρω ότι προέρχεται από τον τομέα των επιχειρήσεων, έχει μεγάλη εμπειρία, ε, θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Για τον κύριο Σάντ βεβαίω θα είναι χαρά μου να συμμετάσχει και αυτό στι συζητήσει. Είναι ο πρώην Πρωθυπουργό τη Μάλτα, έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για το ευρώ ε, και τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Θα συζητήσουμε τον ρόλο του δημόσιου τομέα τον 21ο αιώνα, Το τομέα των μεταφορών και της ενέργειας ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις ε, χρειάζονται κρατικές ενισχύσεις, όμως από την άλλη αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει πρόσχημα ε, για τη σπατάλη δημοσίων δαπανών χωρίς να υπάρχει ζήτηση από τον ιδιωτικό τομέα. Ε, κάποιοι έχουν τα διπλάσια, τα τριπλάσια αεροδρόμια, παραδείγματο χάρη από αυτά που χρειάζονται. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ μαζί σα. Χρειάζεται μια, χρειάζονται εθνικέ αρχέ ανταγωνισμού. Ε, αυτό αποτελεί μέρο τη δημόσια υπηρεσία που πρέπει να παράσχει το κράτο για να υπάρχει ίσως ανταγωνισμό. Με τον συνάδελφο και φίλο τον κύριο Λούνες ε, Προερχόμαστε από παλές, ε, ε, παλαιά ευρωπαϊκά έθνη τα οποία ανοιχτά στο εμπόριο. Ιστορικά είμαστε κατά της κακής διακυβέρνησης και των κακών μορφών σοσιαλισμού. Ε, έτσι, με φυσικότητα θα έλεγα έχουν υπάρξει, έχει υπάρξει συνένεση για το πώς βλέπουμε την τα οικονομικά ζητήματα, οπότε με χαρά θα συνεργαστούμε. Ενδεχομένως να αναφέρουμε πολύ το Google όπως λέτε, ε, ενδεχομένως να πρέπει να προσέξουμε περισσότερα όταν ονοματίζουμε συγκεκριμένες εταιρείες, όμως από το 2013 και μετά σε όλες τις εκθέσεις ανταγωνισμού, ε, το οποίο το έχουν ψηφίσει 600 μέλη, στο κοινοβούλιο έχει μπει το όνομα Google. Ε, υπήρξε αυτή η ανάγκη. Ε, Βεβαίω ε, δεν είναι ωραίο να ονοματίζουμε συγκεκριμένα και να δαχτυλοδείχνουμε εταιρείε και χώρες, αλλά όταν υπάρχει τόσο ευρία πλειοψηφία είναι απαραίτητο. Τώρα, ε, ε, αν τα, οι, οι υπόλοιποι, ε, τα υπόλοιπα μέλη του Κοινοβουλίου δεν συμφωνήσουν να συμπεριλάβουμε την Google, θα το δεχτώ, διότι είμαι δημοκράτης. Ε, και την κυρία Μπερμέχο, ναι, συμφωνώ με τη διαγνώσή σας για αυτά που συμβαίνουν, παραδείγματο χάρη στον τομέα τη ενέργειας. Γιατί δηλαδή να εισάγουμε τόσο πετρέλαιο, τόσο φυσικό αέριο από τρίτε χώρε, να έχουμε δυνατότητε για την ανάπτυξη νέων πηγών ενέργεια στι δικέ μα χώρε. Να σα θυμίσω ότι η Ισπανία, στην Ισπανία, παραδείγματο χάρη, έχουμε 8 φορέ λιγότερε φωτοβολταϊκέ εγκαταστάσει από τη Γερμανία. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή δηλαδή έχει οχταπλάσιε φωτοβολταϊκέ εγκαταστάσει από ό,τι στη χώρα μου την Ισπανία. Ε, γιατί, γιατί υπήρξε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης ε, μικρών επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οικογενειών ακόμα να αναπτύξουν αυτές τις δομές. Και σε κάποιες άλλες χώρες ε, υπάρχει ακόμα προστατευτισμός, ε, υπάρχουν ολιγοπόλια και διαπιστώνουμε ότι τα κράτη-μέλη αυτά έχουν και τις υψηλότερες τιμές ενέργεια τελικά. Ε, και αυτό βεβαίω πλήττει την ανταγωνιστικότητα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και δημιουργεί φτώχεια στι οικογένειε. Να σα δώσω και ένα άλλο στατιστικό στοιχείο. Η πόλη των Βρυξελών, με τον καιρό που βλέπετε εδώ σήμερα, συχνά τον έχουμε αυτόν τον καιρό, πέρυσι ε, εγκατέστησε περισσότερες φωτοβολταϊκές μονάδες από το σύνολο του κράτους της Ισπανίας. Ε, η Ευρώπη λοιπόν ε, παρέχει αυτά τα στοιχεία, τα απίστευτα και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Μπορούμε να συμφωνήσουμε νομίζω από αυτόν και βέβαια αυτό που είπατε για τα ολιγοπόλια σε διάφορου τομείς ε, και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι αγορές ε, θα είναι ανοιχτές ε, για να μπορέσουμε όμως χρόνο να εξασφαλίσουμε και την επιβίωση των γεωργών τα επόμενα χρόνια, ε, θα συνεργαστούμε για να στείλουμε κάποια μηνύματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους Ευρωπαίους πολίτες που καθημερινά μας ρωτούν τι κάνουμε εδώ. Ευχαριστώ. Κύριος Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα τις απόψεις τους σε σχέση με τις προτάσεις, ε, τις, ε, προτάσεις, τις προτάσεις που περιλαμβάνονται ε, για να δημιουργηθούν χρονικές προθεσμίες για έρευνα για λόγους ανταγωνισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτον θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τρεμόσα για την έκθεσή του, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Λάβαμε υπόψη τις παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης Σχετικά με τις προθεσμίες για τις έρευνες αντιτράστη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ίσως να μην είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Έχουμε κάποια μέσα στη διάθεσή μας ήδη, τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να πάρουμε σε έφθετο χρόνο τις αποφάσεις και προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε με τον πιο σωστό τρόπο σαν παράδειγμα τις διαδικασίες αντικαρτέλ, τις οποίες έχουμε, οι οποίες ε, πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε μία διετία. Υπάρχουν και άλλα μέσα τα οποία ε, μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν οι χρονικές προθεσμίες με αποτελεσματικό τρόπο και να καλυφθούν οι ανησυχίες μας. Οι έρευνες οι τομεακές τις οποίες κάνουμε μας επιτρέπουν να συλλέγουμε τις πληροφορίες και τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση μεμονωμένων συγκεκριμένων τομέων. Ταυτόχρονα όμως το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο, οι περιπτώσεις αυτές ε, σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι ιδιαίτερα περίπλοκες και γι' αυτό θα πρέπει να σεβόμαστε τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα σχετικά με τις υπερασπιστικές ε, ε, δυνατότητες των εμπλεκομένων πλευρών. Συνεπώς λοιπόν πιστεύουμε ότι οι χρονικές προθεσμίες όπως τις προτείνεται δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάρουμε σωστές και γρήγορες αποφάσεις. Ένας άλλος τρόπος επιτάχυνσης ε, στη λήψη των αποφάσεων είναι να έχουμε τους απαιτούμενους πόρους και γι' αυτό καλωσορίζουμε σε εισαγωγικά τις ε, προτάσεις μας ως προς αυτό. Ευχαριστούμε και το Κοινοβούλιο διότι πραγματικά ε, πρέπει να ζητήσει και σωστά κάνει την ανεξαρτησία των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, κάτι το οποίο θα βοηθήσει η εσωτερική αγορά να λειτουργήσει σωστά για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Ο εισηγητής πάρα πολύ σύντομα, 30 δευτερόλεπτα μόνο, κατανοώ βέβαια την αυξανόμενη περιπλοκότητα των θεμάτων αντιτράστ. Θα πρέπει όμως να την εξισορροπήσουμε την περιπλοκότητα αυτή με μέτρα χωρίς να περάσουν από την άλλη πλευρά. Οι επιχειρήσεις πρέπει φυσικά έχουν δικαίωμα υπεράσπισης, αλλά δεν μπορεί μια υπόθεση να κρατάει 10 χρόνια. Γιατί καταστρέφεται ο ανταγωνισμός, υποκύπτουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνεχίζονται τα μονοπόλια. Γι' αυτό λοιπόν απαιτείται να υπάρχει μια ισορροπία σαφής η στην οποία αναφερθήκατε αλλά όχι να υπάρχει απεριόριστος χρόνος ε, στις προσπάθειες έβρεσης λύσης. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, το χρονοδιάγραμμα εδώ είναι η προθεσμία κατάθεσης 20 Νοεμβρίου τροπολογιών, εξέταση των τροπολογιών τον Ιανουάριο, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς, θα σας ενημερώσουμε και η ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ τον Φεβρουάριο. και περνάμε στην Ολομέλεια στη συνέχεια, αλλά θα σας ενημερώσουμε και για αυτές τις ημερομηνίε. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή, του Σκιώδης και την Επιτροπή. Τώρα περνάμε στο σημείο 8. 6 και 7, 6 τώρα, δύο γνωμοδοτήσεις. Consider the amendments. Λοιπόν, εγώ ως εισηγητής ε, να πω ότι υπάρχουν δύο τροπολογήσεις, προτάσεις τροπολόγησης σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από πλευράς των κρατών μελών για την άσκηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής ε, των εκτελεστικών της αρμοδιοτήτων. Εγώ είχα πει από τον προηγούμενο μήνα ότι θα καταθέσω την πρότασή μου σχετικά με την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα τροπολογήσει τον κανονισμό για την επιτροπολογία. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεσή μου και τον οποίο ο βασικός στόχος είναι η αύξηση της διαφάνειας. Έχουν κατα, κατατεθεί 10 τροπολογίες. Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που κατέθεσαν τις τροπολογίες αυτές. Στην πλειοψηφία τους ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση θα έλεγα. Η διαφάνεια είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει σεβαστό σε όλα τα επίπεδα και αυτό ισχύει και σε επίπεδο επιτροπής και σε επίπεδο δεύτερης και στο δεύτερο επίπεδο είναι πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κατανοεί τις θέσεις που ακολουθούν τα κράτη-μέλη και επίσης ε, τίθεται και το θέμα της καλύτερης νομοθετικής δραστηριότητας της πρόσβασης στο Μητρό και στις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται. Δεν βλέπω εδώ μαζί μας τον κύριο Έκχαρτ. Έχω κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με τις τροπολογίες 7 και 11 τις οποίες έχει καταθέσει. Τροπολογίες οι οποίες ουσιαστικά θα αφαιρέσουν την ουσία από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρεί ότι εδώ η άποψή μου είναι διαφορετική εντελώς από τη δική του, αλλά φυσικά θέλω να ακούσω και τις ε, απόψεις των συναδέλφων για όλα αυτά. Πρώτος ομιλητής δεν είναι εδώ. Η κυρία Μάλετιτς και γι' αυτό θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο των συντηρητικών. Ευχαριστώ Πρόεδρε και πολύ σύντομα να πω ότι υπάρχουν πολύ λίγες ε, τροπολογίες, ε, ε, δύο από τις οποίες είναι δικές μου, οπότε βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση σας κοινοποιήσω ότι ε, το ECR είναι διατεθειμένο να υποστηρίξει αυτήν την χρήσιμη διαφάνεια που περιλαμβάνεται εδώ. Θα δείτε για παράδειγμα στην τροπολογία μου 16 ότι θέλω να διασφαλίσω ότι η πρόθεση νομοθετική στο πρώτο επίπεδο ε, απηχείται σωστά και στο δεύτερο επίπεδο. Αυτό αυτός είναι ο στόχος αυτής της τροπολογίας. Σε, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες 7 και 11, ε, όπως είπατε και εσείς ε, και εγώ, δεν είμαι βέβαια ότι ε, συμφωνώ με την αξιολόγηση των κανόνων ψηφοφορία των ε, πρασίνων. θεωρώ δηλαδή πως η συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων είναι σημαντική, αλλά θα ήθελα βέβαια να ακούσω και αναμένω να ακούσω την αιτιολόγηση για αυτή την προτινόμενη διαγραφή. Θα περιοριστώ σε αυτά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλοι ομιλητέ. Θα προσπαθήσω προφανώ να έρθω σε επαφή με του συναδέλφου κατά την ε, ε, προετοιμασία των συμβαστικών ε, τροπολογιών. Σα ευχαριστώ για την παρουσίαση που κάνατε μόλι τώρα, συνάδελφοι, των τροπολογιών σα. Τροπολογία 16 συγκεκριμένα. Και εμεί ε, θεωρούμε ότι εδώ δηλαδή η νομική πράξη θα ε, πρέπει να είναι συμβατή με την νομοθεσία και το περιεχόμενο θα πρέπει να πηχεί και την πρόθεσή μα ε, φυσικά. Αλλά Ορισμένε περιπτώσει είναι γνωστέ όπου, για παράδειγμα, υπάρχουν αιτιολογικέ σκέψει όπου δεν καθίσταται σαφέ το τι ακριβώ εννοούμε. Άρα, επί τη αρχή συμφωνούμε μαζί σα ότι πρόκειται εδώ για μια σαφή υποχρέωση η οποία και κατοχυρώνεται και στη συνθήκη. σε ό,τι αφορά δηλαδή τις ανάγκες, ε, τους στόχους και τους περιορισμούς σε ό,τι αφορά τις ε, εξουσίες. Το χρονοδιάγραμμα τώρα. Στι 20 Νοεμβρίου λοιπόν η ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή Έχω και από εκεί και μετά δεν ε, ε, ε, ξέρουμε πότε θα γίνει η ψηφοφορία στην ε, επί της αρμόδια Επιτροπή. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Μία ακόμα γνωμοδότηση. Ε, σε ό,τι αφορά την Αρμενία και την υλοποίηση τη Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση τη νομοθεσία. Ε, Στι 10 ε, Οκτωβρίου που έγινε ε, μια συζήτηση, παρουσίασα το σχέδιο τη νομοθεσία μου για αυτό το ζήτημα και χαίρομαι που κάποιοι από εσά επέδειξαν ενδιαφέρον και υπέβαλαν τροπολογίε. 23 τροπολογίε συνολικά υποβλήθηκαν και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω όλου για ε, τη συμβολή σας προκειμένου να βελτιωθεί αυτή η γνωμοδότηση. Θα πρέπει να σας πω πως η γενική μου ε, αξιολόγηση αυτών των τροπολογιών είναι θετική, καθώς ε, όλες τους υποστηρίζουν τη βασική γραμμή που ακολουθώ σε αυτήν την γνωμοδότηση, που είναι ακριβώς η καλύτερη θεσμική συνεργασία και βελτίωση της νομοθεσίας. Και οι περισσότερες βέβαια από τις ε, τροπολογίες ε, εστιάζουν στην ενίσχυση της θέσης μας ή στην έμφαση, της έμφασης που δίνουμε κάποιες ε, ε, στην άμπλυνση αν θέλετε του χαρακτήρα ε, της νομοδότησης πάντως σε γενικές γραμμές τροπολογίες είναι συμβατές μεταξύ τους οπότε δεν νομίζω πως θα υπάρξει πρόβλημα στο να φτάσουμε σε ένα συμβασμό σε σχέση με αυτές ε, παρόλα αυτά συμφωνώ περισσότερο με κάποιες τροπολογίες, ενώ με άλλες υπάρχει κάποιος, ε, κάποια περιθώρια συζήτησης. Ε, ε, οπότε σε γενικές γραμμές συμφωνώ με αυτές τις τροπολογίες αλλά θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα πώς θα φτάσουμε στον μεγαλύτερο δυνατό, στη μεγαλύτερη δυνατή ομοφωνία σε σχέση με αυτέ. Κύριο Μαρτουσέλο δεν είναι εδώ. κύριο Φόξ θα πάρετε και πάρετε το λόγο, Ναι, και πάλι πολύ σύντομα να σας πω ότι από πλευρά του ΙΣΕΑ μπορούμε να υποστηρίξουμε πολλές από τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της διαφάνειας αλλά και της νομοθετικής συνέχειας μεταξύ επίπεδου 1 και επίπεδου 2 ε, σε ό,τι αφορά τις ε, περαιτέρω ε, παραπομπές που γίνονται, σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις μας, ναι, και αυτό μπορούμε να το υποστηρίξουμε, όπως και την έκκληση του να είναι το Συμβούλιο πιο διαφανές αλλά και ε, τροπολογίες που μας καλούν να λάβουμε περισσότερο υπόψη μας ε, ε, τον τριμερή χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων. Ε, σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο για αυτό το ζήτημα. Άρα μάλλον διμερή είναι η συζήτηση που κάνουμε αυτά τα ζητήματα σήμερα εδώ, παρόλα αυτά χρήσιμη. Και ούτως ή άλλως μια σειρά από τροπολογίες είναι πολύ σαφείς ως προς το τι περιλαμβάνουν. Οπότε θα έρθω σε επαφή με τους ε, συντάκτες αυτών των τοπολογιών για να φτάσουμε σε έναν συμβασμό. Το χρονοδιάγραμμα 21 ε, Νοεμβρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή και δεν ξέρουμε πότε θα λάβει η χώρα η ψηφοφορία της ουσίας αρμόδια Επιτροπή. Τώρα θα περάσουμε στα σημεία 8 και 9. Η οδηγία για το νομικό και υπηρεσιακό πλαίσιο της ηλεκτρονικής κάρτας ευρωπαϊκών υπηρεσιών και ο κανονισμός πάλι για την ηλεκτρονική κάρτα και τις σχετικές ε, διοικητικές διευκολύνσεις. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ είναι εδώ η αρμόδια, αλλά ε, και εμείς νομοδοτούμε. Ο κύριος Λούτφιξον είναι ο εισηγητής μας. Όλε έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις τροπολογίες που, μου έστειλαν. Πολύτιμα όλα αυτά και χρήσιμα. Αλλά βεβαίως ε, υπάρχει και κάποια πόλωση. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Κάποιοι υποστηρίζουν την πρόταση, θέλουν να την κάνουν πιο στεναρή, κάποιοι άλλοι ε, θέλουν απλά να την απορρίψουν. Ε, εγώ θεωρώ, η δική μου μάλλον άποψη για την πρόσθεση της Κομισιόν δεν έχει αλλάξει. Ε, υπάρχει λόγος βεβαίως ε, να έχει κανείς αμφιβολία, να αμφισβητεί τον λόγο ύπαρξης αυτής της πρωτοβουλίας. Υπάρχουν, υπάρχει μεγάλη ε, ασάφεια ό,τι αφορά την άποψη των πολιτικών ομάδων απέναντι στην πρόσθεση τη Κομισιόν και αυτό φαίνεται και στι τροπολογίε. Ε, γι' αυτό λοιπόν έχω και εγώ ε, υποβάλει μια τροπολογία έτσι ώστε να είναι πιο δύσκολο να είναι πιο δύσκολη η φοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή και οι εικονικές εταιρείες οι εταιρείες με εικονική έδρα ε, Είναι σαφές βεβαίως ότι υπάρχει ε, διχασμός και μέσα στις πολιτικές ομάδες απέναντι στην πρόταση της, ε, ε, της Κομισιόν. Πολλοί απορρίπτουν παντελώς την πρόταση της Κομισιόν. Υπάρχει μια άλλη σαφήνειας. θα ήταν καλό να διευκρινιστούν κάποια πράγματα πριν προχωρήσουν οι εργασίες μας. Νομίζω ότι υπάρχει μια κάποια συμφωνία για κάποιους τομείς ε, που παρουσιάζουν πρόβλημα και υπάρχει μια τροπολογία που λέει ότι πρέπει να, υποκλειστεί, να θα αποκλειστεί ο τομέας των κατασκευών. Ο κατασκευαστικός τομέας, πληκτρονική κάρτα. Ε, κάποιες ομάδες θεωρούν ότι αυτή ότι ο χαρακτήρας ε, ε, ο διαχρονικός της κάρτας είναι προβληματικός, αλλά βέβαια αν βάλουμε ένα όριο ε, χρονικό, ποιο θα είναι αυτό το όριο. Ε, δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Η προθεσμία που θα πρέπει να ισχύει για τις εθνικές αρχές να εξετάσουν, να εξετάσουν τα σχετικά αιτήματα είναι πολύ μικρή. Δεν δίνει στα κράτη-μέλη την δυνατότητα να αντιμετωπίσουν σωστά ε, να επεξεργαστούν σωστά τις αιτήσει. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε μια λογική προθεσμία. Πάντως η πρόταση της Κομισιόν προλέπει μια πολύ σφιχτή προθεσμία, γι' αυτό και υπάρχουν πολλές τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή κάποιες από τις προθεσμίες γενικότερα στην πρόταση να αυξηθούν. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ασφάλειες, ε, η Κομισιόν είναι σαφής εδώ. Πολλοί θέλουν να αφαιρέσουμε την ασφάλεια από την πρόταση. Κάποιοι άλλοι θέλουν απλώ να γίνουν κάποιε τροποποιήσει. Θα είναι δύσκολο να συγκεράσουμε τι απόψει, αλλά θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση σε βάθο για όλα αυτά, για να μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή οδό. Τώρα από εκεί και πέρα, να σα ευχαριστήσω, Πρόεδρε, που μου δώσατε το λόγο και αναμένω να ακούσω τι έχουν να πούν και όλοι οι Ευχαριστώ. Να δούμε και ποιοι είναι εδώ όμως για να μιλήσουν, λέει ο πρόεδρος. Φούλβια θα πάρεις το λόγο για την έκθεση του κυρίου Λούτφιξον. E uh, για την ηλεκτρονική κάρτα. Ευχαριστώ. Τον εισηγητή για την προσπάθεια την οποία έκανε. Είναι σημαντικό το πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας και υπάρχουν και αντιφατικές αντιλήψεις γύρω από αυτό. Η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε είναι να εργαστούμε ακόμα περισσότερο για να βελτιώσουμε την πρόταση και να υπάρξει μια σωστά διαφρομένη γνωμοδότηση η οποία να βοηθήσει πράγματι να βρεθεί μια λύση. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ακούσαμε διαφορετικές απόψεις και αναφέρομαι σαν παράδειγμα στην διάρκεια η οποία προς το παρόν προβλέπεται να είναι αόριστη. Υπάρχουν προτάσεις για τριετή διάρκεια που να οδηγεί σε μια ανανέωση για μια περίοδο δεκαετή. Ένα άλλο θέμα είναι ο τομέας των, της οικοδομής. Ο τομέας αυτός είναι ένας από τους βασικούς στόχους και είναι ένας από τους τομείς τους οποίους βρίσκονται τα περισσότερα εμπόδια στον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της Ένωσης αλλά είναι κάτι που ισχύει ίσως και για κάποιους άλλους τομείς βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς. Ελπίζω, εν πάση περιπτώσει, στην επόμενη συνάντηση των σκιωδών να συνεχίσουμε την προσπάθεια Εγώ φυσικά θα σταθώ στην τελική απόφαση την οποία θα πάρουμε με δημοκρατικό τρόπο. Θα υποστηρίξω τη συνέχεια των εργασιών και ελπίζω να καταλήξουμε σε μια σωστή πρόταση. Από το ΕΣΥΑΡ ο Σολζόκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, το ECR το βλέπει θετικά ότι έχουν υποβληθεί 130 τροπολογίες. Ε, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι και τόσο καλή η πρόταση της Κομισιόν. Όμως ε, συχνά οι εκθέσεις της Κομισιόν αφήνουν μεγάλο περιθώριο βελτίωση. Ορισμένε φορέ βέβαια γίνεται να βελτιωθεί, ορισμένε φορές δεν γίνεται καν να βελτιωθεί. Εμείς έχουμε βάλει τροπολογίε ε, ε, για να διευκρινίσουμε του ορισμού. Ε, ε, να αυξήσουμε την νομική ασφάλεια. Μπορεί να προστηρίξουμε και τις προτάσεις άλλων πολιτικών ομάδων που μειώνουν την διάρκεια ισχύω ε, της ηλεκτρονικής κάρτας, να, να υπάρχει δηλαδή κάποιο όριο. Θα μπορούσαμε να δεχτούμε τέσσερα χρόνια, παραδείγματο χάρη. Ε, ε, το οποίο μετά να μπορεί να ανανεωθεί έως και δέκα χρόνια. Αλλά αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες και τους φόβους ε, των χωρών ε, υποδοχής, οπότε μπορούμε να δεχτούμε μια, ένα χρονικό όριο ανώτατο, ε, μια προθεσμία πιο μεγάλη, για να μπορεί να γίνει η επεξεργασία της αίτησης. και για την, οικονομική, την ελάχιστη οικονομική δραστηριότητα και τα ζητήματα ψευτοαυτοαπασχόλησης. πρέπει να το δούμε αυτά. Ε, πάντως οι τροπολογίε θέλουν ακόμα δουλειά. Πολλέ. Ε, ε, ουσιαστικά αμφισβητούν το σύνολο του εγχειρήματο. Ε, να μπορεί ένα κράτο μέλος να αποφασίσει κατά πόσο μπορεί να γίνει αποδεκτή μια εταιρεία ή όχι. Αυτό, τέτοιες τροπολογίες δεν αφήνουν κανένα περιθώριο συμβασμού. Εν πάση περιπτώσει, συνοψίζοντας, ε, εμείς ε, θα υποστηρίξουμε τον εισηγητή ε, στην προσπάθεια βελτίωσης της αφήνειας και της νομικής ασφάλειας του κειμένου σε ό,τι αφορά την ταχύτητα των διαδικασιών και σε ό,τι αφορά τις απειλές, την απάλληψη των απειλών από τις απειλές ψευτοαυτοαπασχολούμενων. Αλλά οι τροπολογίε οι οποίε ε, πραγματικά πλήττουν αυτό το project ε, δεν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε διότι είναι κρίσιμο αυτό το project, αυτό, αυτή η πρωτοβουλία για το μέλλον της ευρωπαϊκής ε, αγοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν, υπάρχει από τους φιλελευθέρου. όχι, εδώ είναι η Παλώμα Βεβέχο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών απαιτεί σωστές συνθήκες και για τους παρόχους και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις και σχέσεις εμπιστοσύνη σε όλα τα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει ε, να πάρει μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην υπάρξει περαιτέρω επιτάχυνση στις προσπάθειες οι οποίες γίνονται για την απορρίθμιση της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει ο κανονισμός το ταχύτερο δυνατόν να εφαρμοστεί. Βλέπουμε στην Ισπανία ότι δεν εφαρμόζεται σωστά σε τομείς όπως ε, οι συγκοινωνίες, οι μεταφορές κτλ. Από την άλλη η ανταλλαγή ε, πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη πάρα πολύ συχνά είναι ε, πολύ βασικές και πολύ απλές μάλλον και δεν δίνουν την δυνατότητα σωστής ενημέρωσης. Η έλλειψη επίσης κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι το σημαντικό για να αποφύγουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ. Δεν μπορεί να μην υπάρχει η δυνατότητα να ανακαλέσει ένα κράτος μέλος τις άδειες παροχής που έχει εκδώσει μια διαφορετική χώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα βοηθήσει στους καταναλωτές και στους πολίτες να πιστέψουν πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό εμείς θα κάνουμε πρόταση απόρριψης της συγκεκριμένης πρότασης. Σας ευχαριστώ. Ένας έχει ζητήσει το λόγο για το κατσάι, η κυρία Περές. Κοιτάξτε, εγώ δεν ήθελα να παρατείνουμε τις συζητήσεις και δεν ζήτησα το λόγο σήμερα σε όλη τη συνεδρίαση, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες τροπολογίες εδώ, οι οποίες τίνουν στην απόρριψη της πρότασης και κάποιες προτάσεις οι οποίες απορρίπτουν τα τμήματα της πρότασης που είναι στις δικές μας αρμοδιότητες, όπως το θέμα των ασφαλιών σαν παράδειγμα. Νομίζω ότι αυτή είναι άλλωστε το κομμάτι, αυτό είναι το κομμάτι της πρότασης το οποίο είναι το πλέον ακατάλληλο. Πριν λοιπόν μπούμε σε μια λογική θα έλεγα συμβιβαστική, να εξετάσουμε σε επίπεδο αρμοδιοτήτων δικών μας το θέμα δηλαδή της ασφάλειας και εγώ θα ήθελα εδώ να ζητήσω από τον εισηγητή μας να μπει μέσα στο θέμα ακριβώς με ξεκάθαρο τρόπο. Γι' αυτό άλλωστε ζητείται και η δική μας άποψη. Για τις ασφάλειες εγώ δεν βλέπω να υπάρχουν αυτή τη στιγμή βιώσιμες σχετικά προτάσεις. Πρέπει να υπενθυμίσω εδώ το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό. Αυτό που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να κάνουμε μία στροφή 180 μοιρών στον τομέα της ασφάλειας σε σχέση με την πολιτική που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα. Αυτό που κάναμε μέχρι τώρα ήταν η εναρμόνιση. Και αυτό το οποίο μας προτείνεται είναι η αμοιβαία αναγνώριση, απλά χωρίς κανένα επίπεδο ισοτιμίας. Συνεπώς λοιπόν νομίζω ότι για τη δική μας πρόταση, για τα θέματα τα οποία μας αφορούν, θα πρέπει να απορρίψουμε το κομμάτι αυτό και κατά συνέπεια νομίζω ότι ε, τα υπόλοιπα θέματα που δεν είναι τμήμα των αρμοδιοτήτων μας δεν θα πρέπει να συζητηθούν ε, πάρα πολύ στο εσωτερικό της Επιτροπής μας. Να τα αφήσουμε στις άλλες, τις αρμόδιες Επιτροπές. Αυτή είναι η άποψή μου τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ. Ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι εύκολο να λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις αποκλίνουσες απόψεις. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να ε, αρκεστούμε στην αρμοδιότητα που έχουμε εμείς στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Η επόμενη συνάντηση των σχεδίων συγκητών τώρα, εκεί θα θέλω να συζητήσω μαζί τους σε βάθο το θέμα. Είναι απαραίτητο. Είναι προφανέ ότι δεν είναι εύκολο να βρεθεί κοινό τόπο. Βεβαίω έχω και εγώ τι απόψει μου. Αναμένουμε με επιμονησία λοιπόν τη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών ε, και θα τα πούμε εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Vote in Econ for November. Ο χρονοδιάγραμμα βλέπει 4 Νοεμβρίου. Δεκεμβρίου, Δεκεμβρίου, συγγνώμη, Δεκεμβρίου, 4 Νοεμβρίου, πέρασε, λέει ο Πρόεδρος, δύσκολο να ψηφίσουμε τον 4 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, η επόμενη συνάντησή μας θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου, στις 23 και συνεχίζουμε και 21 βεβαίως όλη τη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θεός,